Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Και έχουμε φτάσει στα σημεία 9 έως 14 σχετικά με την απαλλαγή. απαλλαγή για τους διάφορους τομείς στους οποίους έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή μας. Και έχουμε την αρμόδια εισηγήτρια που τα έχει εξετάσει όλα. Όλα αυτά για τα οποία είναι αρμόδια από πλευρά τη Επιτροπή Περιβάλλοντο έχουμε την Utah Haug, που παίζει σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή Προπολογισμού και θα της δώσουμε το λόγο για την έκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί όλοι οι συνάδελφοι έχουν λάβει τα έγγραφα, οπότε μπορείτε να τα έχετε διαβάσει. Σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν τα έγγραφα, άρα ξέρετε γιατί πράγμα μιλάμε. αν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι σε κάποιο τμήμα για κάποιον οργανισμό ή ε, στη γενική έκθεση για τον τομέα περιβάλλοντος και υγείας. Ευχαρίστως μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες οι συνάδελφοι. Η προθεσμία έχει τεθεί για 1η Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μέχρι τότε μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις για τα πάντα. Αλλά αν και τώρα έχουν οι συνάδελφοι κάποια πρόταση, μπορείτε να μου κάνετε κάποια υπόδειξη, ευχαρίστω να το ακούσω. Ε, καθώς με αφορά, θέλω να πω ότι ε, όταν τα ετοιμάζουμε εκ των προτέρων, γιατί πρέπει να προβλέψουμε και το χρόνο μετάφρασης και όλα αυτά, ε, μπορεί κάποια σημεία να χρειάζονται κάποια τροποποίηση. Ευχαρίστω λοιπόν να κάνω κάποιες τροποποίησεις αν αυτό απαιτείται. Για το δημοσιονομικό έτο 2008 μπορούμε να πούμε γενικά ότι είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το ποσοστό εκτέλεσης ε, είναι καλό, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία. Για την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος Όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος, η εκτέλεση ανήλθε στο 95,15%. Είχαμε ικανοποιητικό ποσοστό εκτέλεσης λοιπόν για απορρόφηση των μέτρων. Για την δημόσια υγεία φτάσαμε στο 99,75%. Με θαυμασμό το βλέπει κανείς ένα τέτοιο ποσοστό, αλλά φαίνεται όντως έτσι να είναι 99,75% και μένει πολύ μικρό υπόλοιπο ανεκτέλεστο και στον τομέα για την ασφάλεια των τροφίμων και υγεία των ζώων 98%. Πολύ ψηλά ποσοστά, 95, 98, 99,75. Πολύ καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού λοιπόν. Η Επιτροπή εκπροσωπείται εδώ. Έχω δει τουλάχιστον μία εκπρόσωπο της Επιτροπής και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε προς την Επιτροπή ότι έμαθε πια το μάθημά της από τις προηγούμενες φορές και μπορούμε να δώσουμε την απαλλαγή. Έχουμε αρκετά στοιχεία και για την εκτέλεση του προγράμματος live. Η Επιτροπή ε, ήταν πρόθυμη να παρέχει βοήθεια προς τους συμμετέχοντες και έτσι το ποσοστό εκτέλεσης βελτιώθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και στη συνοπτική αιτιολόγηση μου έχω βάλει τα σχετικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται να σας δώσω τώρα όλα ε, τα λεπτομερή στοιχεία. Στο live θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Υπάρχει ένα ορθογραφικό, ένα τυπογραφικό λάθος. Κάπου λέει για τον Ιούλιο 2008 θα έπρεπε να λέει και όχι 2009. Κατά λάθο έχει, έχει μπει σε ένα σημείο ότι δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2009 ενώ θα έπρεπε να πούμε 2008. Αυτά για, το, για την πρώτη ε, γνωμοδότηση, για το γενικό προϋπολογισμό μετά, για τους διάφορους οργανισμούς. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Πολύ ικανοποιητικά στοιχεία όσον αφορά τους διάφορους τομείς. και στην ε, εφαρμογή των μέτρων και στην αξιολόγηση των μέτρων ε, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή είναι το μίσμα με τους οποίους ασχολείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Περιβάλλοντος. Έχει αναλάβει μια λειτουργία επίβλεψης Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, λοιπόν, την ξηρασία, την ερημοποίηση, όλα αυτά είναι δραστηριότητες στις οποίες έχει μια γενική εποπτεία. Και νομίζω ότι όλα τα στοιχεία παρουσιάζονται ικανοποιητικά για το 2008. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, Υπάρχει ίσως μια μικρή καθυστέρηση όσον αφορά τον τομέα της πληροφορικής ε, χρήματα που θα καταβληθούν την επόμενη χρονιά που ε, αυτό αντιβαίνει κάπως στις υποχρεώσεις διατηρήσης του ενιασίου του προϋπολογισμού. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζεται μια μικρή βελτίωση. Το 2009, πάντως, φαίνεται ήδη να έχουν προχωρήσει θετικά τα πράγματα. Όταν θα κάνουμε, λοιπόν, την έκθεση για την απαλλαγή του 2009, ελπίζουμε να μην έχουμε τίποτα να πούμε από αυτού. το προσωπικό που έπρεπε να προσληφθεί προσελήφθη. Και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο, λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε την απαλλαγή. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων, Είχαμε κάποιες δυσκολίες ε, με τη Σουηδία. σχετικά με την έδρα. Ε, φαίνεται να έχουν επιληθεί αυτές οι δυσκολίες. Από, την, από, τον ίδιο τον από το ίδιο το κέντρο πρόληψη και ελέγχου των νόσων, αυτό που ακούμε είναι ότι δεν έχουν όλα επιληθεί, αλλά υπάρχουν θετικά βήματα. Ας μην ενθουσιαστούμε λοιπόν εξ αρχής. Θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με τη Σουηδία για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης και για να τους τονίσουμε το ενδιαφέρον μας. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων είναι το πρώτο επιτυχές έτο, για τον οργανισμό αυτό, το πρώτο επιτυχές έτος. αυτά τα ήταν απαραίτητα για τη δημιουργία και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων ε, έγιναν. Εφαρμόστηκαν αυτά τα οποία έπρεπε να εφαρμοστούν. Έγιναν οι κατάλληλες δαπάνες. Μπορούμε με ικανοποίηση να δηλώσουμε ότι προχωρεί ορθά. και όσον αφορά την οικοδόμηση του κέντρου συνεδριάσεων του οργανισμού, ε, θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια ε, που αναλογούν στον οργανισμό. Και όσον αφορά ε, τον αριθμό των θέσεων προσωπικού, νομίζω ότι έχουν ήδη επιτύχει κατά 95% το στόχο. κάθε εμπειρογνώμων, κάθε ειδικό θα μπορούσε ε, για θέματα χημικών προϊόντων θα μπορούσε να θεωρήσει ως μη ιδανικό τόπο εργασίας στο Ελσίνκι, αλλά κατάφερε αυτός ο οργανισμός ε, χημικών προϊόντων να προσελκύσει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και να συμπληρώσει το 95% του οργανογράμματος. Όσον αφορά την, ε, τον οργανισμό ελέγχου των τροφίμων, δεν έχουμε να πούμε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Έχουν ε, προχωρήσει σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι προς ε, σκέψη, δεν μας απασχολούν, απλώς ε, ε, συνεχίζουμε να τα εξετάζουμε όσον αφορά κάποιο άρθρο που δημοσιεύθηκε για κάποιον που έφυγε από, τον, από την αρχή ελέγχου των τροφίμων και πήγε σε κάποια άλλη εταιρεία. Δεν ισχύει ο ίδιος κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό της αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων όπως ε, για τους υπαλλήλου της Επιτροπής. Πάντως ε, είναι γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητη προσοχή. Δεν είναι όμως θέμα το οποίο ανήκει στην απαλλαγή του 2008. Είχε προταθεί να το συμπεριλάβουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν συνέβη το 2008, συνέβη μετά το 2008, αλλά δεν είναι θέμα που μας απασχολεί τώρα. Υπάρχει μια διοργανική ομάδα εργασίας, ε, Επιτροπή Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ασχολούνται με τους κανονισμούς ε, γενικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προτείνουμε σε αυτή τη διοργανική επιτροπή να εξετάσουν κάποια τέτοια πιθανά θέματα. Θα πρέπει να το σκεφτούν λοιπόν αν χρειάζεται να έχουν ε, τον ίδιο κώδικα διοντολογία σε όλους τους οργανισμούς, ε, τον ίδιο κώδικα που έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να παραιτηθεί κάποιο από την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τρόφιμων και να πάει σε μια φαρμακευτική εταιρεία που ασχολείται με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αλλά όπως σας είπα αυτό δεν είναι θέμα της απαλλαγής του 2008. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους που με βοήθησαν και αυτά δεν είχα να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ τη Γιούτα Χάουγκ. Και ευχαριστούμε γιατί ε, ασχολήθηκε η συντάκτη της νομοδότησης με πολλούς οργανισμούς, με πολλούς τομείς. Είναι ενδιαφέρον ε, μια συνάδελφος που να ασχολείται με τις δαπάνες να λέει ότι καλώς δαπανήθηκαν. Η κυρία Χάουγκ. Ε, εμάς μας ενδιαφέρει ε, να δαπανώνται τα χρήματα για τους στόχους που προβλέπονται. Εμείς ε, θέλουμε να μην δαπανούνται ε, για ε, περιτούς λόγους, καλύτερα να γυρίζουν στα ταμεία των, των χωρών μας. Όταν μένουν υπόλοιπα χρήματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάλι για το καλό. Τόμας Ούλμα βλέπω ότι έχω ζητήσει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και συγχαρητήρια προς τη Γιούτα Χάουγκ, ε, την ευχαριστούμε, γιατί πολύ σωστά προετοίμασε τις γνωμοδοτήσεις. Καταλαβαίνω ότι όταν επιστρέφονται χρήματα στους εθνικούς προϋπολογισμούς μπορεί να χαίρονται οι υπουργοί οι αρμόδιοι για τα οικονομικά σε κάθε χώρα. Πάντως πιστεύω ότι οι γνωμοδοτήσεις είναι ισορροπημένες και είναι καλό το ότι έχουμε υψηλό ποσοστό εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το 90% και 100% είναι πολύ καλά ποσοστά. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία είχαν προγραμματιστεί. Κάποια υπόλοιπα όσον αφορά τον τομέα της πληροφορικής υπάρχουν για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. και για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων. Πίσω ότι είναι θετική ενασχόληση με διάφορες έρευνες θετικό και το ότι λύνονται τα προβλήματα του Κέντρου Πρόληψης Νόσων με την ε, Σουηδική Κυβέρνηση σχετικά με την έδρα. Και ίσως ε, σας κάνω κάποιες προτάσεις ε, για τροπολογίες, για κάποιες λεπτομέρειες. Πάντως γενικά είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ρεμπαντή. Όχι. Η κυρία Λεωτάρ, εάν την πετύχω, συνεχίζοντας τον κατάλογό μου. Η κυρία Χάουγκ. να περιμένουμε τροπολογίες από το ΕΛΚ, από τον κύριο Ούλμα Και αν δεν έχει κανείς άλλο σχόλιο, τι να σας πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ θα υποβάλω δύο-τρεις τροπολογίες για να εκφράζω σαφέστερα αυτό το οποίο δεν έχουμε ίσως εκφράσει επειδή κάναμε πολύ νωρίς την νομοδοτήση. Κυρία Κλάς. Έχω μια ερώτηση σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών ε, Προϊόντων. Είχαμε πει ότι υπάρχουν ε, ε, πολλά τα οποία περιμένουν προς αξιολόγηση σε σχέση με την οδηγία REACH ε, και τώρα βλέπουμε ότι ε, έχουμε υψηλό ποσοστό εκτέλεση του προϋπολογισμού άρα να θεωρήσουμε ότι ε, θα προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα οι εργασίες και δεν θα έχουμε καθυστέρηση στα διάφορα θέματα και σιγά σιγά θα πρέπει να αναλάβει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων περισσότερε εργασίε, περισσότερε δραστηριότητε και για τα βιοκτώνα και για τα παρασιτοκτώνα. Υπάρχουν πολλά τα οποία προ το παρόν λείπουν και θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερη συνεργασία. και θα προσπαθήσω και μαζί με τη Utah Hawk το 5%, ε, του προσωπικού που δεν έχει προσληφθεί ακόμη να φροντίσουμε ε, να καλυφθούν οι θέσεις αυτές για να μπορέσουν να δουλέψουν όσο δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κυρία Χάουγκ, να απαντήσω κατευθείαν στην Κρίστα Κλάς. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέει. Όμως τώρα είμαστε στο 2010 και μιλάμε για τον προϋπολογισμό του 2008. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε. πρέπει να μιλήσουμε τώρα για τον προπολογισμό του 2011. Και νομίζω όταν θα κάνουμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2011 θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό που ζήτησε η Κρίστα Κλάς. Όταν θα μιλάμε λοιπόν για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την επόμενη χρονιά, να κάνουμε αυτές τις προτάσεις ε, στα σχόλιά μας. γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το 2008 ως έτος αναφοράς για να κάνουμε τα σχόλιά μας για το τι δεν κάνουν σωστά τώρα. Σύμφωνα με τη διαδικασία του προϋπολογισμού, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2011 για να κάνουμε τα σχόλια και να ασκήσουμε κάποια πίεση, όπως εννοεί και η Κρίστα. Άννα Ρόσπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι απολύτω ικανοποιημένη. Απλώ θέλω να ρωτήσω την Πρόεδρο. Τι γίνεται με, τον οργανισμό στην Ιρλανδία για τα κτηνιατρικά ζητήματα. Ποια θα είναι η θέση του μέσα σε όλο αυτό το φάσμα οργανισμών. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα σχετικά. Μιλώ για το κτηνιατρικό οργανισμό. Jetzt äh, Χάουγκα, Οργανισμός για τα κτηνιατρικά προϊόντα είναι ένας εκτελεστικός οργανισμός που συνδέεται άμεσα με την Επιτροπή. Δεν είναι δηλαδή αποκεντρωμένος οργανισμός. Δεν οφείλουμε να τους δώσουμε εμείς απαλλαγή λοιπόν. Η Επιτροπή Γεωργίας μπορεί να ασχοληθεί με μια απαλλαγή για αυτά τα θέματα. Οι οργανισμοί σχετικά με τον πολιτισμό και την ε, παιδεία ε, δεν χρειάζονται απαλλαγή από εμά. Εμείς ε, δίνουμε απαλλαγή σε αποκεντρωμένους, όπως αποκαλούνται, οργανισμοί. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσετε την Επιτροπή Γεωργίας πώς προχωρούν σε σχέση με αυτό τον οργανισμό στο Δουβλίνο. Ευχαριστούμε. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 1η Φεβρουαρίου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 23 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας. Να περάσουμε τώρα στην παρουσίαση της κυρίας Ρόσπαχ για το θέμα της ε, προστασίας των ακτών και των υδάτων στο, στην περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού και σε σχέση με ό,τι αφορά τα προβλήματα ρήπανσης ιδιαίτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα είναι αρκετά εύκολο να το παρουσιάσω, είναι σύντομα τα στοιχεία που διαθέτω εδώ. Εδώ έχουμε ρήπανση από πλαστικά στον βορειοανατολικό Ατλαντικό με ένα εμβαδό 20.000 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε για εγκαταλελειμμένα δίχτυα από σκάφη τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πια και όλα αυτά συντελούν στη ρήπανση του βορειοανατολικού Ατλαντικού. Μιλάμε για ένα πρόβλημα αρκετά σημαντικό και εδώ είναι επίσης πήγον να εγκριθεί το πρωτόκολλο. Όπως ε, ξέρετε η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ήδη υπογραφεί, αλλά μόλις το 2008 μπορέσαμε να δώσουμε ένα τέλος στις εδαφικές διαφορές και διεκδικήσεις Ισπανίας-Μαρόκου. Το, το πρωτόκολλο λοιπόν αυτό, το πρόσθετο πρωτόκολλο θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε ακόμα καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι κατάλληλη στιγμή για να αναλάβουμε δράση. Ήδη πέρυσι είχαμε σχολιάσει το θέμα όταν ε, συζητήσαμε το θέμα της κατακράτησης διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ όμως ε, είναι ακόμη πιο σημαντικό το πρόσθετο πρωτόκολλο για τις θάλασσές μας, για την ε, θάλασσα του Βερίγγιου Πορθμού, για τις ακτές της Αφρικής ακόμη. Εδώ μιλάμε για θέματα που απασχολούν τόσο τα, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα υδατά τους, όσο και τρίτες χώρες. Επαναλαμβάνω λοιπόν το ζήτημα είναι σοβαρό. Για να καταπολεμήσουμε τις περιπτώσεις ρήπανσης, το θέμα το συζητάμε έτσι κι αλλιώς από καιρό. Έχουμε τη συμφωνία της, του Ελσίνκη, της Βόνης, τώρα υπάρχει ήδη η συνθήκη της Λισαβόνας που μας επιτρέπει να αναλάβουμε δράση. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι παράκτιες χώρες του Ατλαντικού να κυρώσουν το πρωτόκολλο ώστε να καταπολεμήσουν από κοινού τα σοβαρά ατυχήματα, τα θαλάσσια ατυχήματα. Είτε πρόκειται για περιπτώσεις ε, χημικής ρήπανσης, είτε για πετρελοκυλίδες. Θα πρέπει εδώ να επιδιώξουμε την προστασία των θαλασσίων ειδών, των ψαριών. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνούν όλοι για την κύρωση αυτού του πρόσθετου πρωτοκόλλου προκειμένου να καταπολεμήσουμε προβλήματα της θάλασσας που μας απασχολούν όλο και περισσότερα. Θα παραμείνω σε αυτά τα σχόλια διότι δεν έχω πραγματικά πολλές λεπτομέρειες να σας δώσω. διότι προφανώς ε, τα προβλήματα του κόσμου, του χώρου της θάλασσας δεν σταματούν σε εθνικά σύνορα. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζουν σύνορα και μπορούν να απαντηθούν σε όλες τις περιοχές της υδρογείου. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κυρία Ρόσπα για την εξαιρετική έκθεση. Ο κύριος Ασένης, ο σκοδής εισηγητής μας, έχει κάτι να προσθέσει. Η κυρία Γκέρλινγκ, παρακαλώ. Το Chris Davis. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζουμε την έκθεση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ήταν σε κρεμότητα αρκετά χρόνια και θεωρώ ότι ήγηκε η ώρα να ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπε η συγγήτρια για το θέμα των πλαστικών αποβλήτων, τις τεράστιες ποσότητες που έχουμε στις θάλασσες. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο οποίος είναι σε θέση να απαντήσει. Το θέμα έχει τεθεί στην ημερήσια διάταξη. ποιο είναι ο αρμόδιος ε, στο Συμβούλιο. Ε, υπάρχουν πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, αντιμετώπιση της απόρριψης πλαστικών και άλλων απορριμμάτων από ευρωπαϊκά σκάφη, απόβλητα και σκαφών τρίτων χωρών στι θάλασσε δεν ξέρω αν κάποιος είναι σε θέση καν να απαντήσει. Ε, μήπως, κοιτάξτε προς τα εκεί, προς την Κομισιόν και αν δείτε κάποιον ο οποίος είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει. Αυτό και θα κάνω. Κύριε Αντελανουά, έχετε κάτι να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστούμε, αλλά ανάψτε και το μικροφόνο σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή τη για την θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου αυτού, τη συμφωνία μάλλον. Η συμφωνία επιτέλους 20 χρόνια μετά την υπογραφή της θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα της έκτασης των πλαστικών απορρίτων, της πλαστικής σούπας όπως λέγεται εντό εισαγωγικών, το πρόβλημα αυτό ξεκίνησε στον ειρηνικό. Τα παράκτια κράτη άρχισαν να αναλαμβάνουν δράση για να αντιμετωπίσουν το θέμα. Αλλά για τον Ατλαντικό ωκεανό το φαινόμενο και πρόβλημα επισημάνθηκε από την Ολλανδική Αντιπροσωπεία σε, ένα πρόσφατο, σε μια πρόσφατη σύνοδο του Συμβουλίου και η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν έρευνες για τη μελέτη του ζητήματος. Στην περίπτωση που σε κάποιες γεωγραφικές ζώνες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ε, υδατολογικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα, θα πρέπει να ληφθεί συγκεκριμένη δράση. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληροφόρηση και θα πρέπει να ξεκινήσουν οι σχετικέ έρευνε για αυτό το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την σύμβαση πιο συγκεκριμένα, που θα μπορούσε να καλύψει το πρόβλημα αυτό, αναφέρθηκε η σύμβαση ΟΣΠΑ για την προστασία του βορειοανατολικού Ατλαντικού και πράγματι η πλαστική αυτή σούπα εντό εισαγωγικών θα μπορούσε να καταπολεμηθεί εντό αυτού του πλαισίου. Υπάρχει και η σύμβαση του 1972 για την καταπολέμηση τη θαλάσσια ρήπανση, γνωστή ω Σύμβαση του Λονδίνου. Εδώ λοιπόν συμμεριζόμαστε τις, ε, τη μέρημνα του, της εισηγήτριας και θα δούμε πώς τα διάφορα φόρουμ και περιφερειακές συμφωνίες μπορούν να μας ενισχύσουν στην καταπολέμηση του προβλήματος αυτού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Θα ήθελα λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Ρώση. Ευχαριστώ. Ήρθα λίγο καθυστερημένος, αλλά θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες της εισηγήτριας. Η άποψή μας είναι ευνοϊκή. Την ευχαριστώ για τη δουλειά της. Σας ευχαριστώ όλους. Θα σας παρακαλέσω τώρα να πάρετε τις κάρτες ψηφοφορίας. Σας έχουμε δύο ψηφοφορίες. Η πρώτη για την έκθεση, το σχέδιο απόφασης μάλλον του Συμβουλίου. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Εψήφισαν όλοι με την ένωσή σα. Έχουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι στην Ολομέλεια. Εψήφισαν όλοι. Ναι, λήξη. 24 φαίνεται να ψήφισαν. 24 ψήφοι υπέρ, 0 κατά. Εγκρίθηκε ομόφωνα λοιπόν το σχέδιο απόφαση. Δεύτερη απόφαση τώρα. Σχέδιο ψηφίσματο του Κοινοβουλίου. Να ξαναψηφίσουμε λοιπόν. Έναρξη της ψηφοφορίας. Εψήφισαν όλοι. Λήξη. Και πάλι ωραία ομοφωνία των 24 ψήφων. Σας ευχαριστώ. Κυρία εισηγήτρια, τα συγχαρητήριά μας. Εγκρίνεται ομόφωνα η έκθεση. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και με ιδιαίτερη χαρά θα ακούσουμε τον κύριο Πρόντι για το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Λευκή βίβλος προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Νομίζω ότι στο σημερινό πλαίσιο θα σας ακούσουμε με ιδιαίτερη ενδιαφέρον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Γι' αυτό λοιπόν για κάποια πράγματα θα ήθελα να σας παραπέμψω και στη συνοδευτική δήλωση της ε, συζήτησης που είχαμε την προηγούμενη φορά η Λευκή Βίβλος ήταν πολύ αναμενόμενη, η οποία ε, ξεκινά τη συζήτηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της αλλαγής του κλίματος και υπήρχαν και μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες ολεάνα και αυξάνονταν, ε, καθώς υπήρχαν και άλλες πρωτοβουλίες και άλλοι άξονες, οι οποίοι μας έδιναν κάποια αποτελέσματα, τα οποία ήταν απογοητευτικά, για να μην παραβλέπουμε την τελευταία διάσκεψη της Κοπενχάγης. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει ε, να δούμε ε, στην πράξη πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τα σχέδια και η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή τη λευκή βίβλο δεν κάνει και γιγάντια ε, άλματα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Πρόκειται, όπως έγραψα και στην έκθεσή μου, για ένα προπαρασκευαστικό έργο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εκπονήσουμε στο μέλλον τη βασική στρατηγική και τα βασικά σχέδια δράσης μας. Από αυτή την οπτική γωνία το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλά διαρθρωμένο, ίσως υπάρχουν και κάποια κενά, τα οποία σημαίνει και η έκθεση Επιτροπής Μεταφορών για τις ορεινές περιοχές, για τα μέτρα τα οποία πρέπει να υιοθετήσουμε για να ε, προστατεύσουμε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός και επίσης όπως ε, έχω πει επανειλημμένως, η αλλαγή θα είναι πλήρης και θα αφορά όλες τις πτυχές της ζωής μας, τόσο της εργασιακής όσο και της ιδιωτικής. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ε, ατέρμονο εγχειρίδιο με μέτρα, αλλά μπορούμε να βρούμε μια-δυο άγουσες οι οποίες από εκεί και πέρα θα υιοθετηθούν, θα αποφασιστούν και θα ε, διαχειριστούμε σε τοπικό επίπεδο με μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι λογικό να πούμε ότι κάποιες περιοχές θα πληχθούν περισσότερο από άλλες από την αλλαγή του κλίματος. Ε, δεν μιλάμε πλέον για μετριασμό των αποτελεσμάτων, αλλά για το πώς θα είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και πολύ σημαντικές αλλαγές της θερμοκρασίας, διότι το πρόβλημα θα είναι σοβαρό για όλους και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τα γεωργικά συστήματα, τα βιομηχανικά συστήματα, τις τουριστικές δραστηριότητες, άλλο στα ε, βουνά, άλλο στα δάση, άλλο στις πόλεις, άλλο στην εξοχή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι από κοινού. Να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές ε, ε, πλαίσιο για μέτρων, ε, να προσαρμοστούμε, να έχουμε δεδομένα, να έχουμε μοντέλα, να έχουμε κατάλληλη εποπτεία και να υπάρχει και μία πιο μεγάλη επικοινωνία για το κοινό εν γέννη, αλλά και κυρίως για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια ώστε τα θέματα της προσαρμογής ε, στην αλλαγή του κλίματος να είναι παρόντα σε όλες τις πολιτικές της κυβέρνησης, να έχουμε μια καλύτερη διακυβέρνηση, ακριβώς επειδή η προσαρμογή θα έχει μια πολύ σημαντική εδαφική συνιστόσα, μια συνιστόσα η οποία θα πρέπει να είναι λειτουργική και δεν θα πρέπει να είναι ένας κενός κατάλογος καλών προθέσεων. Το θέμα της ε, ε, χρονική συγκυρία δεν έχει ακόμα ε, λυθεί. Στη Λευκή Βίβλο λέμε ότι δεν θα μπορέσουμε να μιλάμε για σχέδιο δράσης μετά από το, πριν από το 2013. Πρόκειται για κάποιο μακρινό χρονικό ορίζοντα και φαίνεται ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ε, αντιμετωπίσουμε αμέσως τα θέματα των κατεπηγόντων ε, να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και να έχουμε και τις γνώσεις για το μέλλον μας. Στην πραγματικότητα τα χρονικά περιθώρια μόλις μας αρκούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επαγρυπνούμε, ώστε όλα όσα πρέπει να γίνουν να ολοκληρωθούν στα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί. Και Αντίστοιχα, αντίστοιχο σκεπτικό πρέπει να έχουμε και για τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τα έσοδα, τους τρόπους, τον τρόπο κατανομής αρμοδιοτήτων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των τοπικών αρχών. Αυτό το επαναλαμβάνουμε. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλεφθεί και ένα τμήμα των κονδυλίων στο σύστημα ανταλλαγής εκπομπών για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό ε, έγινε ήδη, υπήρξε μια πρώτη δόση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν ε, σύντο, μικρό το ποσό. Και στην έκθεσή μου αναφέρομαι και στη σημασία του νερού, του ύδατος, διότι όλα αυτά είναι συστημικές πτυχές τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε συλλογικά. Κυρίως όσον αφορά στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, τις οποίες θα πρέπει να τις συνδέσουμε και με την ε, ε, προστασία του εδάφους μας. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε και τις πολιτικές για τη δημόσια υγεία, την ε, διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Όλα αυτά είναι στοιχεία στα οποία υπάρχουν επιπτώσεις και θα πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Θα ήθελα εδώ να κάνω κάποιες τελικές ε, σκέψεις η Επιτροπή για το Περιβάλλον της Κοπενχάγης θα πρέπει να έχει συντονιστικό ρόλο ε, στο λεγόμενο μηχανισμό του Clearing House και θα πρέπει επίσης στο μέλλον να προβλέψουμε και ένα συντονιστικό ρόλο ε, στα μέτρα προσαρμογής μέσω ενός συγκεκριμένου οργανισμού είτε στο εσωτερικό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ή μέσω της δημιουργίας ε, μιας ad hoc υπηρεσίας. Επίσης ε, μπορεί να έχει και η διευθυντική ομάδα που ε, έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ως προϋπόθεση να είναι παρόντα και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συμμετέχουν. Ε, προβλέπεται και μια προθεσμία για τις τροπολογίες στις 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 16 Μαρτίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Υπάρχουν και άλλες επιτροπές οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν επί του θέματος, η ΑΦΕΤ, η ΝΤΕΒΕ, η Επιτροπή Απασχόλησης, η ΙΤΡΕ, η ΤΡΑΝ, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι οποίες ε, κάποιες από αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει. Έχουμε επίσης την Άγκρη και τη Γιούρη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους ε, παρακαλώ να λάβουν υπόψη τους όλα όσα έχω διευκρινίσει στην αρχή ότι πρόκειται δηλαδή για ένα έγγραφο το οποίο είναι πριν από τη στρατηγική και δεν θεωρείται μια τελική νομοθετική πράξη, τουλάχιστον όχι ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόντι για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σκυλακάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μερικές βασικές σκέψεις. Καταρχήν, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η κλιματική αλλαγή την οποία θα ζήσουμε στα επόμενα 30, 20 με 30 χρόνια είναι αναπότρεπτη. Οτιδήποτε δηλαδή και να κάνουμε στο επίπεδο της, αντιμε... μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, στο mitigation, θα συμβεί η κλιματική αλλαγή για διάφορους λόγους που όλοι οι δήμονες γνωρίζουν. Η προσαρμογή λοιπόν έχει σημασία επί πολλά χρόνια χαράχθηκε μια πολιτική, μια στρατηγική για την κλιματική αλλαγή που βασιζόταν στην υποβάθμιση της προσαρμογής. Ο λόγος ήταν να μην παρεμποδίσουμε τους στόχους της πρόληψης, η οποία είναι ασφαλώς προτιμότερη. Όμως μια πολιτική που είχε νόημα το 2000, το 1990 δεν έχει το ίδιο νόημα το 2010 και ασφαλώς δεν έχει νόημα το 2020 ή το 2030 όταν οι επιπτώσεις πια θα γίνονται πολύ πιο ε, θα αντιληπτές και στην Ήπειρό μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε η πολιτική της υποβάθμισης της προσαρμογής αντίκειται και στη βασική αρχή της περιβαλλοντικής πολιτικής που είναι ο πληρώνει. Αν έχουμε αρχίσει να έχουμε ζημιές πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουμε για αυτές. Τώρα, βασικό εμπόδιο στην πολιτική προσαρμογής είναι η αβεβαιότητα του φαινομένου, ιδιαίτερα όταν μεταβαίνουμε από το πλανητικό στο περιφερειακό, το εθνικό ή το τοπικό επίπεδο. Δεν μπορούμε ακόμη με επαρκή τρόπο να ταυτίσουμε τα συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα, ένα κυκλώνα ή ένα ζεστό καλοκαίρι, με τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική προσαρμογής θα πρέπει να δώσει έμφαση στην πρόληψη και σε περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι ήδη προφανές. Επί του προκειμένου κειμένου τώρα της Επιτροπής και της εισήγησης του συναδέλφου του κυρίου Πρόντι. Συμφωνώ καταρχήν στο γενικό περιεχόμενο. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ανάγκη για ορισμένες σημαντικές προσθήκες. Πρέπει να ζητήσουμε και είναι ανάγκη να υπάρξει μια πιο καθαρή εικόνα από την Επιτροπή για τις προτεραιότητες ό,τι αφορά την προσαρμογή. Οι συνέπειες του φαινομένου που είναι πιθανόν αναπότρεπτες και θα αρχίσουν να συμβαίνουν, ήδη άρχισαν, προηγούνται. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής ό,τι φορά την προσαρμογή με τον ίδιο τρόπο αν θα συμβούν 60 χρόνια μετά ή 80 χρόνια μετά και αν συμβαίνουν σήμερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε την όξυση των προβλημάτων των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μεσογείου, όπως επίσης και την είσοδο ξένων ειδών, που ήδη συμβαίνουν, ειδικά στις θάλασσες στη Μεσογείου. Είναι πιθανότατα ότι αυτές οι επιπτώσεις σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές. Θα έπρεπε κάπως να προηγούνται σε σχέση, για παράδειγμα, με τις επιπτώσεις ανόδου της θάλασσας που θα έρθουν 70 ή 80 χρόνια μετά με σημαντικό βαθμό. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, εκτός από τις προβλέψεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του κοινοτικού προϋπολογισμού, που είναι όπως ξέρουμε όλοι περιορισμένες, υπάρχουν και τα χρήματα για αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών που είναι περισσότερο αδύνατα και τα οποία προβλέπεται στο ETS, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρήπων, ότι θα δοθούν για mitigation και adaptation, για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Με βάση τη σχετική οδηγία μιλάμε για το 10% του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρήπων. Πιστεύω ότι τα χρήματα αυτά που θα είναι στο μάκρος του χρόνου σημαντικά είναι σωστό να μοιραστούν ισότιμα μεταξύ μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου mitigation και προσαρμογής adaptation. Και σε ό,τι αφορά την προσαρμογή να εισάγουμε την αρχή της προτεραιότητας στις περιοχές και χώρες που θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή, ειδικά στα επόμενα 30 χρόνια, δεν θα έχει ομοιόμορφες επιπτώσεις θα υπάρξουν περιοχές της Ευρώπης που θα πληγούν δυσανάλογα πολύ και άλλες που θα πληγούν ελάχιστα ή καθόλου. Δεν μπορεί τα χρήματα για προσαρμογή να πάνε ομοιόμορφα. Άλλωστε, η βασική αρχή νομικά κατοχυρωμένη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας πολιτικής μας είναι η αρχή του οριπένων πληρώνει. Εδώ ζητούμε η αρχή αυτή να εφαρμοστεί εντός της Ένωσης μόνο για το 5% των εσόδων από τους ρηπαίνοντες. Πρόκειται για το ελάχιστο δυνατό ποσοστό. Τώρα, στα ειδικότερα θέματα για να τελειώσω, πιστεύω ότι πρέπει να περιλάβουμε, εκτός από αυτών που καλύπτονται, ειδικέ αναφορές καταρχήν για τα δάση, εξήγησα γιατί, δεύτερον για τις επιπτώσεις στη βιοπικιλότητα από την μετανάστευση ξένων ειδών, τρίτον για τις επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον, στο αστικό περιβάλλον επισημαίνω ότι λόγω του συνδυασμού του φαινομένου της θερμικής νησίδας που πολλαπλασιάζει στον αστικό χώρο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ανάγκη να μας απασχολήσει ειδικότερα το τι θα συμβαίνει στις πόλεις διότι υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής εκεί, η θερμική νησίδα. Τέταρτον, η επιπτώση στην οικονομική δραστηριότητα που πρέπει να αποτελούν ένα χωριστό κεφάλαιο. Και τέλος, οι επιπτώσεις από τα πιθανά νέα μεταναστευτικά ρεύματα που θα προκληθούν, μια που ξέρουμε ότι οι βασικές πηγές μετανάστευσης, η Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία, για την Ευρώπη, θα είναι ε, περιοχές που κατεξοχήν θα πληγούν από τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Je, je je remercie. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα θα αλλάξω ιδιότητα για δύο λεπτά για να αναλάβω αυτήν τη σκιώδους εισηγήτρια για την έκθεση του κυρίου Πρόντι. σα ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόντι για τη δουλειά σα. και να πω ότι συμμερίζομαι απολύτω μαζί σα τι ανησυχίε σα. για το γεγονό ότι αυτή η λευκή βίβλος δεν αποδίδει τον κατεπίδο χαρακτήρα που θέλαμε στην αντιμετώπιση τη πρόκληση. Έχουμε συζητήσει διαμακρών για τι κλιματικέ αλλαγέ. προετοιμάζουμε πολλά και ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγέ διότι προφανώς μας αφορά άμεσα. Επηρεάζεται η καθημερινότητά μας, η παραγωγή και η κατανάλωσή μας. Και γι' αυτό ίσως και να δυσκολευόμαστε. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα συμπεριληφθούν οι κοινοτικές πολιτικές στους στόχους της προσαρμογής και πώς θα τους επιδιώξουμε τους στόχους αυτούς. Η λευκή δίβλωση είναι ένας τρόπος να δώσουμε έμφαση στην ατεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των ε, συστημάτων της φύσης και εδώ βλέπουμε την ε, δυνατότητα συνεργασίας και την δοκιμασία του πόσο μπορούν να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές συνεχείς. Εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόντι για τη σημασία που δίνει σε μια οδηγία πλαίσιο για τα εδάφη. Η κατακράτηση του διοξιδίου του άνθρακα, η προστασία από πλημμύρε, η προστασία από τη διάβρωση, η καλή κατάσταση των οικοσυστημάτων, η αγροτική παραγωγικότητα, όλα αυτά εξαρτώνται άμεσα από τη δυνατότητά μα, τη δική μα, να προστατεύσουμε και να ανανεώσουμε, να αναζωογονήσουμε τα ευρωπαϊκά εδάφη η, ίδια η κατάσταση της γης θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά μας να μεταρρυθμίσουμε τις ε, γεωργικές μας πρακτικές ώστε να γίνουν πραγματικά βιώσιμες. Υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσε η έκθεση να αναφέρει τη σημασία της βιοποικιλότητας, της προώθησης της γεωργικής βιοποικιλότητας, διότι αυτή είναι μια προϋπόθεση για την προσαρμογή μας. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας για τον, ε, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, εδώ αυτό ο παράγοντα είναι καθοριστικό, ιδίω σε σχέση με τι μεταβολέ τη θερμοκρασία, όπου τα θαλάσσια οικοσυστήματα επηρεάζονται ούτω ή άλλω ιδιαίτερα από τι ανθρωπογενεί δραστηριότητε, κυρίω την υπεραλίευση. Χρειάζεται ταχεία εφαρμογή τη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και βεβαίω κάποιες, κάποια στοιχεία κλειδιά, μέτρα κλειδιά για να μπορέσουν να αντισταθούν τα οικοσυστήματα. Επίσης είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε τις γνώσεις μας. Δεδομένης της σημασίας του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου των κλιματικών αλλαγών χρειάζονται μέθοδοι συμμετοχής ε, σε έρευνες όπως το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας για τις επιστημονικές δραστηριότητες, το ονομαζόμενο επιστήμη και κοινωνία που επέτρεψε την, ε, το σχεδιασμό στοχευμένων ενεργειών, τη συνεργασία των τοπικών παραγόντων και την καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Τέλος, εφόσον πρέπει να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας, να μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε αρκετές γνώσεις στην κατοχή μας για να μην αναβάλουμε περαιτέρω τη δράση μας. Κυρία Πρόντι, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας για τον καταπήγοντα χαρακτήρα της ε, δράσης που πρέπει να αναλυθεί εδώ. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον στο παρελθόν είχαμε μια πραγματική στρατηγική προσαρμογή και αναλόγως και τώρα να ε, πορευτούμε. Ευχαριστώ. Λόγω στον κύριο Μπασακούτα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Πρόντου για αυτό το πρώτο σχέδιο έκθεσης. Ε, πρόκειται για πάρα πολύ καλό κείμενο και μάλιστα διευκρινίζει και κάποια σημεία στα οποία είναι ασαφής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε όλοι ε, τα θέματα τα οποία άπτονται της αλλαγής του κλίματος και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα στη Λευκή Βίβλο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σαφής τι σημαίνει, ως προς το τι σημαίνει αυτό για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και νομίζω ότι ο κύριος Πρόντι πολύ καλά επισημαίνει κάποια από αυτά τα σημεία. Θα ήθελα να προσθέσω προσθέσω κι εγώ κάποια βέβαια. Ε, Καταρχά, η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα από τα βασικά μέτρα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ η ερώτησή μου είναι η εξή. Καλύπτει την προσαρμογή σε αυτό το στάδιο και έχει εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τούδε κατά πόσον αυτές οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, ασχολούνται παρκώς με το θέμα της προσαρμογής του κλίματος και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό και στην απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, η προσαρμογή στην γεωργική πολιτική. Αυτό είναι ένα από τους βασικούς άξονες. Εδώ νομίζω μπορούμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, διότι αν μιλάμε για την ε, ε, μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική, η αλλαγή του κλίματο θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των μεταρρυθμίσεων τη κοινή αγροτική πολιτική. Και νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο θέμα χωρί να είναι πάρα πολύ σαφή για το τι ακριβώ εννοούμε. Και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για γεωργία και επιδοτήσει στη γεωργία, θα πρέπει ίσω να ε, πληρώνουμε περισσότερο για υπηρεσίε οικοσυστημάτων και να δούμε θέματα βιοποικιλότητα, προστασία του του εδάφους, ε, οικολογικές δραστηριότητες, ε, μορφολογία του εδάφους, όλα αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε όταν μιλάμε για κοινή αγροτική πολιτική και μεταρρυθμισή της. Τώρα, η διασύνδεση με την υγεία και τις κοινωνικές πολιτικές. Ε, το θέμα των ασθενειών των ζώων δεν αντιμετωπίζεται σωστά στη Λευκή Βίβλο. Η διασύνδεση με τις ασθένειες ζώων θα πρέπει να διευκρινιστεί. Και μια συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Πρόντι για το σημείο 17 όπου μιλά για την ε, συμμετοχή των ασφαλιστικών βιομηχανιών. Τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Είναι πιο συγκεκριμένη ερώτηση προς τον εισηγητή λοιπόν αυτή. Για το θέμα της βιοποκυλότητας, όπως ε, αναφέρατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα να επισημάνω ότι αν μιλάμε για χρηματοδότηση του Natura 2000, δεν είναι αρμόδια μόνο τα κρατομέλη για τη χρηματοδότηση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει το λιθαράκι της, να δει και αυτή λίγο τα θέματα της χρηματοδότησης και νομίζω ότι και η βασική ερώτηση εν τέλει είναι σε ποιο βαθμό χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσέγγιση για την προσαρμογή του κλίματος θα πρέπει να είμαστε λίγο περισσότερο σαφείς. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση και να είμαστε λίγο πιο σαφείς και να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε μία οδηγία στην οποία τα κράτη-μέλη ναι μεν θα κάνουν και αυτά τη δουλειά της, αλλά χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή οδηγία για την προσαρμογή. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς από αυτό. Εν κατακλείδη, αν μιλάμε για προσαρμογή του κλίματος και τη Λευκή Βίβλο, ε, όλα αφορούν την επόμενη τριετία. Μιλάμε για μια μακροπρόθεσμη διαπραγμάτευση που θα σχετίζεται φυσικά και με τη συζήτηση για τον προπολογισμό που θα γίνει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Αλλά νομίζω ότι κάποια θέματα χρήζουν άμεση αντιμετώπιση γιατί η αλλαγή του κλίματο ήδη συμβαίνει, επομένω πρέπει να ετοιμαστούμε. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι στα τρέχοντα προγράμματα οικονομικής ανάκτησης, ανάκαμψης υπάρχουν ε, και κάποια πράγματα για την αλλαγή του κλίματος. επομένω θα πρέπει να δούμε και την προσαρμογή στο κλίμα και να μην την αναβάλουμε τη συζήτηση για την επόμενη τριετία. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πάλι να πω ότι είναι έξοχη η έκθεσή σα, κύριε Πρόντι, απλώ πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι από ό,τι ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή τη Βίβλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλαναν. Ίσως να πάρω εγώ το λόγο στη θέση του κύριου Κάλαναν, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Εκ μέρους της ίδιας ομάδας ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πρόντι και εγώ. Νομίζω ότι και εμείς, λίγο πολύ σαν τους προηγούμενους ομιλητές, συμφωνούμε ότι μιλάμε για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και μετριασμό των συνεπειών τους εδώ και κάποιο καιρό, αλλά φαίνεται να δυσκολευόμαστε να την υλοποιήσουμε αυτή την προσαρμογή. Συμφωνώ λοιπόν ότι αυτά που προτείνει η Λευκή Βιβλός για την προσαρμογή δεν επαρκούν. Δεν είναι συγκεκριμένα τα μέτρα που προτείνονται και οι προτάσεις. Μετά τη σύνοδο της Κοπενχάγης είδαμε, και είναι και ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αμέσω μετά, ότι υπήρξαν δηλώσεις για την προσαρμογή, αλλά δεν υπήρξε κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στο μέλλον, τις ε, προσεχείς εβδομάδες και μήνες και το πρόγραμμα της προσαρμογής θα πρέπει κάπως να το συμπληρώσουμε με συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε. Πριν δώσουμε το λόγο στον επόμενο αγορητή, απλώς να σας πω ότι στην αίθουσα έχουμε μια, ένα τηλεοπτικό δίκτυο εκ μέρους του ΕΛΚ. Φαντάζομαι να μην υπάρχει αντίρρηση. Για λόγους διαφάνειας απλώς οφείλω να σας το επισημάνω. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόντι, όπως και οι προλαλήσαντες, για το σχέδιο κειμένου που μας παρουσίασε σήμερα. Νομίζω ότι αρχίζει πλέον να δίνει σάρκα και οστά σε αυτό που πρέπει να περιλαμβάνεται στην Λευκή Βίβλο και να ζητάει και λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, διότι τις χρειαζόμαστε. Πρέπει να είμαστε πιο διεξοδικοί. Κάποιος ανέφερε πριν όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά γενικώ πρέπει να δούμε και το 2020 και την όλη στρατηγική που προσπαθεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς βλέπει τα επόμενα βήματα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετά σαφή τα πράγματα. Και από τη Λευκή Βίβλο δεν προκύπτει πού ακριβώς θα το βάλουμε αυτό στην ε, όλη αυτή διαδικασία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η προσαρμογή και ο μετριασμός θα βρίσκονται στο επίκεντρο. για το πώς βλέπουμε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης για τις ε, μελλοντικές μας πολιτικές. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε τη δήλωσή μας εμείς. Ε, δεν είναι μόνο θέμα χρηματοδότηση. Οι παράγραφοι 26 και 27 πρέπει να περιλαμβάνουν κάποιες πιο σαφείς δηλώσεις για το πώς θα πρέπει να είναι η όλη διαδικασία και το όλο θέμα της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής θα πρέπει να βρίσκεται στον επόμενο γύρο χρηματοδοτήσεων. Έχουμε και ένα κατάλογο επιτροπών οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ευρύ είναι το φάσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών που ε, θεωρούμε ότι ε, θα επηρεαστούν από την προσαρμογή τα θέματα του προπολογισμού, η γεωργία, η περιφερειακή ανάπτυξη και το πόσο σημαντικά είναι αυτά. Συμφωνώ με όλα όσα ακούσαμε για τα θέματα της βιοποικιλότητας. Υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα επιδράσει αυτό στο θέμα των δικαιωμάτων, στο θέμα του ύδατος για παράδειγμα. Είναι απλώς θέμα πόρων ή είναι και το δικαίωμα στην πρόσβαση σε νερό. Και επίσης ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Κάποιοι αναφέρθηκαν στους ανθρώπους που θα έρθουν στις ακτές μας τι θα γίνει με όλους αυτούς οι οποίοι θα γίνουν πρόσφυγες λόγω του κλίματος. Στο παρελθόν στην Επιτροπή μας έχουμε συζητήσει και νομίζω ότι αυτό θα προκύψει και στη συζήτηση για την Κοπενχάγη και το τι γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόση βοήθεια πρέπει να δοθεί στις πιο ευάλωτες και φτωχότερες χώρες. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται εδώ σε όλα όσα λέμε και στην έκθεση πώς ε, η Λευκή Βίβλος ε, σε θέματα προσαρμογής θα τα συμπεριλάβει αυτά. Ο κύριος Πρόντι σαφέστατα λέει ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα των εσόδων των κρατών μελών και τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά πρέπει να επισημάνουμε και την ανάγκη στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, να βοηθήσουμε τις φτωχότερες και τις πιο ευάλωτες. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόντι για τα όσα μας είπε και προσβλέπω και στις περαιτέρω συζητήσεις. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ήθελα να επισημάνω σήμερα, αλλά υπάρχουν και κάποιες πάρα πολύ καλές παρατηρήσεις που έγιναν από άλλους συναδέλφους. Ευχαριστούμε κυρία Δεμπρέν. Η κυρία Ρόσπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και οι προλαλήσαντες, και εγώ πιστεύω ότι εδώ πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην προσέγγιση μας. Στη Λευκή Βίβλο γίνεται πολλή λόγος για αναλύσεις, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου πρακτικά στοιχεία, δεδομένα και προτάσεις. Εδώ θα να δοθεί έμφαση στο νερό, διότι όπως γνωρίζετε, χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Λέγεται εδώ ότι θα έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις. Αυτό σίγουρα ισχύει ήδη για κάποιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σε άλλες, αντιθέτως, έχουμε πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις από ό,τι συνήθως. βροχή, χιόνι και ούτω καθεξής. Γιατί λοιπόν δεν προτείνεται κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει λόγου χάρη να δούμε τι γίνεται με τον νότο της Ευρώπης, όπου θα θέλαμε να βρέχει περισσότερο, υπάρχει και το πρόβλημα της αποψήλωση των δασών. Ενώ στο βορρά έχουμε φράγματα και πολλές φορές πυκνό δίκτυο φραγμάτων ή έχουμε την ε, πλοήγηση των ποταμών και μόλις βρέξει λίγο λιγότερο καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Ή οι πλημμύρες. Οι πλημμύρες στην Πολωνία τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μου τα διάφορα κράτη της Ένωσης να σχεδιάσουν κοινά προγράμματα ώστε από κοινού να διαχειριστούν το στοιχείο αυτό, να φροντίσουν να έχουμε κάτι συγκεκριμένο, κάτι ρεαλιστικό στα χέρια μας για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε την κυρία Ρόσμπαχ. Ο κύριος Ασένης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντω έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την υφόρο ανάπτυξη. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον Βιτόριο για αυτή τη θαυμάσια έκθεση. Είναι ένα από τους λίγους ανθρώπους ε, που έχει τόσο ξεκάθαρη εικόνα και γνώση του θέματος τη προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και θα ήθελα να τονίσω και κάποια θέματα που έχουν σχέση με τη βιοπικιλότητα. Είναι σημαντικό Επίσης, να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική όσον αφορά τα δάση της, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. να λάβουμε υπόψη όλα τα θέματα, ε, το πλαίσιο για την προστασία της θάλασσας, ε, για τους οικοτόπους, για την προστασία των πτηνών, να συνδέσουμε όλα αυτά τα θέματα για τα προστατευόμενα διατήματα και νομίζω ότι όλα αυτά είναι προτεραιότητε στον τομέα τη προσαρμογή. Επίση, ε, υποστηρίζουμε την πρόταση τη Επιτροπή για τι κατευθυντήριε γραμμέ σχετικά με την ε, κλιματική αλλαγή και τι περιοχέ Natura. Πολύ σημαντικό είναι. θα πρέπει η προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή να ε, περάσει σε όλες τις πολιτικές ε, και στα θέματα ασφάλειας και στα θέματα περιβάλλοντος και στα θέματα ανάπτυξης. Είναι μια πολιτική εξουσιαστική σημαντική για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλα τα άλλα σημεία του κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει αυτή η πολιτική να μπει και σε όλα τα θέματα εμπορίου, διεθνών διαπραγματεύσεων κλπ. θα πρέπει να έχουμε και στρατηγικές προσαρμογής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και συμφωνώ με το σχόλιο του κυρίου Σκυλακάκη ότι, υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες προσαρμογής σε διάφορες περιφέρειες της ευρωπαϊκή Ένωσης που πρέπει να οδηγήσουν σε διαφορετικό επίπεδο χρηματοδότησης για κάθε περιφέρεια. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι ότι τώρα όλοι οι οικονομικοί φορείς λειτουργούν σαν να μην υπάρχει το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι διάφορες βιομηχανίες, οι διάφοροι κλάδοι, η φαρμακοβιομηχανία διαπραγματεύονται σαν να βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ενώ θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να περάσουν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την οικονομία, τους πόρους και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για να αξιολογήσουμε διαφορετικά σενάρια προσαρμογής και να αποτελέσει και τη βάση του κοινωνικού διαλόγου. Τέλος, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία και τη βασική νομοθεσία σε τομείς ανταγωνισμού υπό το φως της ανάγκης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και να μην δίδονται συγκεκαλυμμένες επιδοτήσεις σε τομείς ε, της οικονομίας που δεν το αξίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη μιλήτρια, κυρία Μακάβεν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα απλώ να συγχαρώ τον Βιτόριο Πρόντι για την έκθεσή του. Είναι πολύ καλή. Υπάρχει όριο στον αριθμό των λέξεων που μπορεί να φτάσει μια έκθεση και κατάφερε να συμπεριλάβει ε, όλα τα σημαντικά σημεία. Είναι μια πρώτη παρουσίαση και οι λεπτομέρειες θα μπουν αργότερα όσο μπαίνουμε στην περίοδο προγραμματισμού. Το θέμα των δημοσιονομικών προοπτικών είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προ το Βιτόριο ή προ την Επιτροπή. Όταν υποβάλλονται προτάσει για την πολιτική ελεία ή για την γεωργική πολιτική, γίνεται αυτομάτως και κάποια αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτάσεων αυτών για την κλιματική αλλαγή. Και ο Κρήτον Αρσένη ε, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό το mainstreaming και στι εμπορικέ πολιτικέ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έννοια της επίπτωσης στην κλιματική αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Μπορεί να ακούγεται γραφειοκρατικό, αλλά όταν θεωρούμε ότι πρέπει να βάλουμε τη σφραγίδα του ότι έχουν εξεταστεί επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, μας κάνει να σκεφτόμαστε κάθε μέτρο με ιδιαίτερο τρόπο. Και κάτι που θα μπορούσαμε να προτείνουμε στη γενική εισαγωγή είναι κάτι για τα ωφέλη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης θέσης εργασίας και είναι και κομμάτι ε, της στρατηγικής για το 2020 τεράστια ωφέλη για την προσαρμογή των υποδομών μας και του τρόπου ζωής μας. Μια μικρή τροποποίηση λοιπόν σε αυτό το σημείο θα τη θέλαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία Grazie. Ευχαριστώ. Καταρχάς, στην έκθεση του κυρίου Πρόντι σημειώνω το γεγονός ότι εκφράζει την εκτίμησή του προς την Λευκή Βίβλο εντελώς αντίθετα με τα όσα είχαμε ψηφίσει στην ε, Επιτροπή μας, διότι σε αυτό το ψήφισμα, το οποίο αμφισβητήσαμε εμείς, έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει η ίδια τις αναδυόμενες χώρες, ε, να αναλάβει το βάρος της αύξησης ε, του ποσοστού της μείωσης των εκπομπών ανεξάρτητα από το ε, ποσοστό στο οποίο θα είχαμε συμφωνήσει. Φαίνεται όμως ότι προσγειωθήκαμε πλέον γιατί και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, ο Γιώ Λάινεν, ήθελε ένα κείμενο το οποίο από εκεί και πέρα ε, στο, ε, στη διάσκεψη των 15 θεωρήθηκε ανύπαρκτο. Ενώ τώρα επιστρέφουμε στη Λευκή Βίβλο, η οποία αναφέρεται σαφώς ε, στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και του φαινομένου του θερμοκηπίου. Λέμε ότι θα πρέπει να το μειώσουμε κατά 15% σε σχέση με τις τιμές του 1990 ε, και αυτό θα πρέπει να γίνει και σε περίπτωση συμφωνίας διεθνούς που δεσμεύει τις βιομηχανοποιημένες χώρες να κάνουν αντίστοιχες μειώσεις. Οι πιο οικονομικά προηγμένες χώρες θα πρέπει ε, να δράσουν ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ευθύνες τους. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο είχαμε ε, προτάξει ω αντίρρηση στο ψήφισμα που ε, εγκρίναμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με χαροποιεί λοιπόν ιδιαίτερο το γεγονός ότι ο κύριος Πρόντι ε, προτιμά τη Λευκή Βίβλο και εγκρίνει τη Λευκή Βίβλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να κάνω τώρα δύο παρατηρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται και στη Λευκή Βίβλο και στο κείμενο του κυρίου Πρόντι και είναι ε, τα ποσοστά ATS. Εμείς δεν είμαστε κατά σε μια τέτοια διάταξη, σε μια τέτοια πρωτοβουλία, ούτε καν στο γεγονός ότι μέρος των εσόδων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μειωθούν οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο θα μπορούσε ίσως να γίνει βορρά στα θηρία και σε κάποια χρόνια να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην οικονομία. Διότι όταν λέμε ότι θέλουμε να συνδέσουμε χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία μπορεί να είναι πηγές επενδύσεων, μπορεί να είναι ομόλογα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, με πακέτα καπνού, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ουσιαστικά μας φαίνεται επικίνδυνο. Δεν λέμε όχι, λέμε απλώς να βρούμε μία λύση και να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεύρει την κατάλληλη λύση προκειμένου να υπήρχε πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος για όλους όσους θα διαχειριστούν τις εκπομπές, το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS. Θα πρέπει να έχουμε ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα το οποίο από εκεί και πέρα θα προσφέρει διασφαλίσεις και στα κρατη και σε όλους όσους θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Εδώ να πω επίσης ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε λίγο, όπως έλεγε και η συνάδελφες Ρόσμπαχ, ε, τα όσα λέει η Λευκή Βίβλος. Δεν είναι αλήθεια ότι έχουν μειωθεί οι βροχοπτώσεις. Μπορεί να άλλαξε το σύστημα της βροχόπτωσης ή της χιονόπτωσης. Έχουμε μεγάλες ποσότητες βροχοπτήσεων σε κάποιες περιοχές και μικρότερες ποσότητες βροχή σε άλλες. Αλλά η συνολική ποσότητα βροχόπτωσης στην Ευρώπη, από τα στοιχεία που έχω εγώ, έχει αυξηθεί, δεν έχει μειωθεί. Φυσικά είναι καταστρεπτικά τα αποτελέσματα, διότι πέφτει με διαφορετικό τρόπο η βροχή από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Επομένω και εδώ είναι καλύτερο αυτό που λέει ο ε, συνάδελφο Πρόντι σε σχέση με αυτό που γράφεται στη Λευκή Βίβλο. Μία τελευταία παρατήρηση ε, την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως είναι η εξή Στην αιτιολογική έκθεση και είμαι πάντα στην έκθεση του ε, Βιτόριο Πρόντι να του ζητήσω το εξή. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί καμιά φορά γράφονται πράγματα τα οποία μπορεί να παρερμηνευθούν. Εμεί έχουμε ζήσει πλημμύρε στην Ευρώπη, αλλά έχουν υπάρξει πλημμύρε και σε όλη την. Ε, στην Ιταλία, συγγνώμη, και έχουν υπάρξει πλημμύρε και σε όλη την Ευρώπη. Ορισμένε φορέ, επειδή υπήρχε υπερβολική βροχό περίπτωση σε μικρό χρονικό διάστημα τα ποτάμια μας δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού και εδώ αναφέρομαι στην Ιταλία πολλά ποτάμια, ε, πολλές γέφυρες συγγνώμη, καταστράφηκαν και αναγκαστήκαμε να κατασκευάσουμε μεγαλύτερες για να μπορέσει να περάσει το νερό. Εδώ λέμε ότι θα πρέπει να ε, έχουμε τη δυνατότητα τα ύδατα να, να κάνουν μεγαλύτερη κρατα... κράτηση. Αυτό θα ήταν λογικό εάν η βροχόπτωση ήταν ομαλή και δεν ήταν υπερβολική. Αν έχουμε όμως πλημμύρα και υπερβολική βροχόπτωση, αν έχουμε δημιουργήσει δυνατότητες μεγαλύτερης κατακράτησης, θα δημιουργηθούν προβλήματα και θα υπάρχουν προβλήματα ακόμα μεγαλύτερα από αυτά που διαπιστώθηκαν στο παρελθόν. Συμφωνώ Εάν καταφέρουμε όταν έχουμε μικρό, λιγότερο νερό να το διατηρήσουμε στις πορείες των υδάτων θα ήταν πολύ καλό. Αλλά όταν βρέχει πάρα πολύ και ήδη έχει πλημμυρίσει το ποτάμι, αν έχουμε δώσει τη δυνατότητα στο ποτάμι να κάνει μεγαλύτερη κατακράτηση, επομένως να καθυστερήσει η ροή του, θα δημιουργήσουμε ακόμα πιο καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. αλλά είναι απαραίτητες ε, οι είναι απαραίτητες ε, οι προβλέψεις για πιθανές πλημμύρες, γιατί αν βρέχει πολύ χρειάζονται κάποιες ε, προηγούμενες ρυθμίσεις για να αποφύγουμε τις καταστροφές. Κύριε Σακλάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο πρώτη για την έκθεσή του. Είναι πολύ καλό αυτό το οποίο μιλάει για τη δημιουργία μιας γνωστικής ε, βάσης, ε, γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά και πρέπει ε, να ενημερώσουμε, θα πρέπει να προσφέρουμε γνώση, να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία για να προχωρήσουμε προς μεγαλύτερη σταθερότητα και στο θέμα της συζήτηση για το κλίμα. Να συνδυάσουμε αυτά τα οποία έχουμε στην έρευνα, στην ανάπτυξη και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα της καινοτομίας, γιατί έτσι προστατεύουμε καλύτερα τους πόρους μας. Το θέμα της γεωργίας αναφέρεται σε δύο σημεία και συμφωνώ με αυτό που είπε η Λίντα Μακάβεν. Είναι πολύ σημαντικό και εδώ να έχουμε ένα σημείο, ένα μέσο αντικειμενικού υπολογισμού. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική βάση όπως είπαμε και να έχουμε ένα μοντέλο υπολογισμού γιατί ε, και στη γεωργία υπάρχουν, υπάρχει και το output και το input. Να γίνεται λοιπόν ένα συνολικός υπολογισμός. Δεν έχουμε μέχρι τώρα κανένα σαφή επιστημονικό υπολογισμό. Να μην υπερβάλλουμε στα μέτρα τα οποία θα λαμβάνουμε, αλλά να έχουμε ε, ακριβή επιστημονικά δεδομένα για να μπορούμε να κρίνουμε και για το θέμα του εδάφους ε, έχει βάλει ο συνάδελφος πρώτη ένα σημείο μόνο. Ίσως είναι πολύ σύντομη αυτή η παράγραφος. Ε, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια οδηγία για το έδαφος και για την προστασία του εδάφους. Ξέρω ότι δεν συμφωνούμε όλοι για το ίδιο θέμα, για το τι ακριβώς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε μια τέτοια οδηγία και αν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα επ' αυτού. Θα διαφωνήσουμε επί των γενικών αρχών επ' αυτού και για την βασική αρμοδιότητα. Τα κράτη-μέλη έχουν τη βασική αρμοδιότητα για την προστασία του εδάφου και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι στον τομέα των υποδομών για το έδαφο υπάρχει ευθύνη των κρατών μελών για τη συντήρηση και την προστασία του εδάφους για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Σε αυτό το σημείο λοιπόν για το έδαφος θα έπρεπε κάπως διαφορετικά να βρούμε την κατάλληλη σύνταξη. Και έχει σχέση και με τις υποδομές το θέμα του εδάφους. Αλλά γενικά πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι πολύ καλή. Προωθεί αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρίχαρτ Ζέιμπερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Βιτόριο Πρόντι, επιστήμονας άνθρωπος, έκανε μια πολύ καλή έκθεση και η Λευκή Βίβλος θα πρέπει να θεωρείται ως Λευκή Βίβλος που θα αποτελέσει βάση συζητήσεων. Υπάρχουν πολλά άλλα, πολύ πιο συγκεκριμένα που μπορούμε από εκεί για πέρα να συζητήσουμε. Αλλά αυτό, αυτή τη Λευκή Βίβλο μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για τη συζήτηση. Ε, συζητήθηκε το θέμα των συμπληρωματικών επιστημονικών δεδομένων που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει ε, να έχουμε τα τελευταία δεδομένα για την αξιολόγηση, δεδομένα δορυφόρων κλπ. Αυτά, ε, όπως είπε και ο συνάδελφος Ορέστε ε, Ρώση, αυτά είναι θέματα επιστημονικά για τα, για οποία υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες και σε επιστημονικό επίπεδο και είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε και τις υδρολογικές επιπτώσεις. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά δεδομένα και να μπορέσουμε εμείς να καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατές συγκεκριμένες προτάσεις. Και η χώρα που εκπέμπει τις, τα περισσότερα, τα μεγαλύτερες ποσότητες ε, η Κίνα είναι μια χώρα για την οποία θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα. Φαίνεται ότι δεν είναι αδιαμφισβήτητα επιστημονικά τα δεδομένα τα οποία δίνει η Κίνα για τις εκπομπές της. Θέλουμε να περιορίσουμε λοιπόν τις εκπομπές, ιδίως από τις χώρες που έχουν τις υψηλότερες εκπομπές, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, και γι' αυτό ακριβώς μας χρειάζονται αυτά τα δεδομένα. Και να παρακαλέσω τον Βιτόριο να συμπεριλάβει και κάτι ακόμη για τα μέτρα κλιματικής αλλαγής. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι θέματα που βρίσκονται στη διεπαφή διαφόρων τομέων. Δηλαδή αυτά τα οποία γίνονται στον ένα τομέα σαφώς έχουν επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Και οι διάφοροι άλλοι τομείς έχουν επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν ε, ε, ε, ακριβώς να συνδέσουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε όλους τους τομείς. Και όσον αφορά τους ε, αμφισβητούντες στην, τα θέματα της κλιματικής ε, ε, αλλαγής, αν σκεφτούμε ε, τον πληθυσμό της γης το 2050, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πόροι μας πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αποτελεσματικό και για τους πόρους ε, και για, την, ε, για τα ορυκτά καύσιμα και για όλες τις πηγές ενέργειας. Θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει ότι θέλει να παραμείνει στο προσκήνιο, να παραμείνει πρώτη μεταξύ όλων των χωρών και γι' αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε και τα θέματα της επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μην έχουμε μακροπρόθεσμα προβλήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουν λεφθεί τόσα για αυτή τη λευκή βίβλο και την έκθεση βεβαίως που σχετικώ μα υποβλήθη από τον κύριο Πρόντι που πραγματικά βρίσκω ότι είναι απολύτως εύστοχο να αναζητούμε τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Πολλά μάλιστα προτείνονται ήδη από τον κύριο Πρόντι, πολλές διαφορετικές μορφές μέτρων και όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα αλλά έχω παρόλα αυτά μια ανησυχία. Όταν βλέπουμε πόσο δυσκολευόμαστε με την οδηγία για τα εδάφη, για τη γη και το πόσο έχει μπλοκαριστεί η οδηγία αυτή στο επίπεδο του Συμβουλίου. Διερωτώ τα μέτρα που προτείνονται και θα προκύψουν από αυτή τη Λευκή Δίβλο και αφορούν τα σχέδια του χωροταξίας των πόλεων, τις άδειες οικοδόμησης, και τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε πολύ διαφορετικούς τομείς. Εδώ νομίζω ότι κάθε φορά θα προσκρούμε στην ε, διάθεση και τη βούληση του Συμβουλίου. Με το χαρακτηριστικό παράδειγμα της οδηγίας ΣΟΛ για τα εδάφη. Δεν ξέρω κατά πόσον δεν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι χρειάζεται και αιμονή, ε, επιμονή μάλλον, για να μπορέσουμε στην υλοποίηση των ε, διευθυντικών ταμείων να συμπεριλάβουμε την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Ίσως αυτό είναι το μόνο μέσο για να επιβάλλουμε με κάποιο τρόπο στο Συμβούλιο την υποχρέωση να λάβει υπόψη ότι πρέπει να προβλεφθούν μέτρα για προσαρμογές στις κλιματικές αλλαγές. Εάν εν τέλει στα διαφορετικά ταμεία πούμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα προσαρμογής, ίσως και να επηρεάσουμε το Συμβούλιο, να αναγκάσουμε να κινηθεί ώστε να λάβει υπόψη και να αποδεχτεί οδηγίες όπως αυτές που σχετίζονται με την έκθεση του κυρίου Πρόντι. Βλέπουμε το τέλμα στο οποίο έχουμε περιέλθει με το Συμβούλιο στο, στην οδηγία αυτή. Ξέρουμε πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουμε. Ενώ πρέπει να ψηφιστούν οδηγίες που θα επηρεάσουν τον ρόλο των τοπικά εκλεγμένων και των πολιτικών ανδρών και γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, σε αυτό ήθελα να σταθώ, γιατί έχουμε πολύ ωραίες ιδέες, αλλά έπειτα όταν θέλουμε να τις κάνουμε πράξη, συναντούμε πολλές δυσκολίες, ιδίως με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Merci. Karin Kadenbach. Herzlichen Dank. Auch ich möchte... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Και θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο στα σημεία το σημείο 4 να συμπεριλάβουμε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και θα επιτύχουμε στον τομέα της προστασίας του κλίματος ε, ε, μόνο αν έχουμε τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Να υπάρχει λοιπόν και μια συνοδευτική εκστρατεία πληροφόρησης και παράλληλα με την υλοποίηση των μέτρων να, μπορεί, να μπορούν οι πολίτες ε, να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης με την κατάλληλη εκπαίδευση, με την κατάλληλη ευαισθητοποίηση και ιδίω στους νέους από την αρχή μέσα στην εκπαίδευση να ενταχθούν τέτοια θέματα. Επίσης, είναι κάτι το οποίο ο συνάδελφος πρώτη το έχει βάλει στο κεφάλαιο υποδομή, ενώ εγώ θα το βάζα στα θέματα μεταφορών και κινητικότητας, ε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάποια πρόοδο στον τομέα της μεταφοράς και των μεταφορών και τη κινητικότητας για να μπορέσουμε να έχουμε στο μέλλον αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον ε, καθηγητά Πρόντι για όλο το έργο που έχει επιτελέσει ως τώρα και βεβαίως όλους τους συναδέλφους σας για την συζήτηση, τα σχόλια, τις συνεισφορές τους. Μεγέρθησαν πολλά ζητήματα εδώ. Θα προσπαθήσω λοιπόν και εγώ να σχολιάσω κάποια από τα σημαντικότερα κατά την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα η ευρωπαϊκή διάσταση της προσαρμογής. Η Λευκή Διβλός αναγνωρίζει ότι περισσότερες από τις δράσεις για τον αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών αποφασίζονται αναπερίπτωση και σε τοπικό επίπεδο. Πολλά από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν λοιπόν πρέπει να ληφθούν ακριβώς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο υπάρχει μια ξεκάθαρα ευρωπαϊκή διάσταση σε όλα αυτά. Το πώς θα χειριστούμε δηλαδή το σχεδιασμό των μέτρων, διότι ο αντίκτυπος ε, των αλλαγών, ιδίως στα νερά, στη βιοπικιλότητα. Είναι σαφώς διασυνοριακά ζητήματα. Υπάρχει εδώ ένα θέμα αλληλεγγύης μεταξύ των περιφερειών. Την ε, ασυμμετρική, τη δυσανάλογη δηλαδή κατανομή των ε, συνεπειών. Η Γεωργία είναι ένας τομέας ιδιαίτερα ολοκληρωμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι αλλαγές στη διοικητική διαχείριση, στους κανονισμούς, θα πρέπει να οριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προφανώς. Δεν μπορεί το κάθε κράτο να έχει απλώ το δικό του μεμονωμένο σύστημα. Και έπειτα τίθεται και το σύστημα τη ε, κερδοφορία, τη αποτελεσματικότητα ω προ το κόστο και τη έρευνα καθώ και τη βάση τη θεμελίωση όλων αυτών ε, των θεμάτων στη γνώση. Δεν μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να τα κατακαιρματίσουμε σε 27 κράτη-μέλη και σε 27 ξεχωριστές δράσεις. Τώρα, η μελέτη αντικτύπου. Υπάρχουν επιπτώσεις στο καθιστός των υδάτων, στη βιοπικιλότητα, στη χρήση των γεών. Και υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Υπάρχουν σημεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, των ε, ε, συστημάτων των υδάτινων και για, ακριβώς να πετύχουμε αποτελεσματική προστασία από τις, τις μενείς επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Ιδίω όπου το κόστο τίνει να διωγγώνεται σε σχέση με την οικοδόμηση υποδομών. Εκεί θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η Λευκή Βίβλος υπογραμμίζει ότι υπάρχουν κενά στι γνώσει μα. Ήδη δεν γνωρίζουμε λίγα βεβαίω, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να μάθουμε. Βασίζεται λοιπόν η Λευκή Βίβλος στην ιδέα ότι πρέπει να αναλάβουμε δράσει τώρα, εκεί που μπορούμε, γιατί έχουμε βεβαιότητα για το τι κάνουμε. Διαθέτουμε ήδη κάποια εργαλεία στα χέρια μα. Έχουμε μια οδηγία για τις πλημμύρες λόγω χάρη, όπου ανατίθεται στα κράτη-μέλη να οργανώσουν προγράμματα για την προστασία από τις πλημμύρες. Ίσως αυτό να, μην είναι το μόνο που θα μας σώσει, αλλά είναι ήδη κάτι. Υπάρχει επίσης, υπάρχουν μέτρα χρηματοδότησης περιφερειακής, γεωργικής, για σκοπούς προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Περαιτέρω μέτρα μπορεί να αναλυθούν για την αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων, της άρδευσης, της καλλιεργήσιμης γης, και όλα αυτά και σε επίπεδο εθνική πολιτική, εφόσον τα κράτη-μέλη δώσουν έμφαση σε αυτά στη δική τους, ε, στα πλαίσια τη δική του ανάπτυξη τη υπαίθρου, λόγου χάρη. Τώρα υπάρχουν τομεί στου οποίου βεβαίω μα λείπουν στοιχεία και χρειάζεται συνολικότερη παρόλα αυτά δράση. Αυτά θα πρέπει να τα αποφασίσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον καλύψουμε όλα τα κενά στις γνώσει μα. Γι' αυτό το σκοπό λέμε ότι χρειάζεται μια σφαιρική συνολική στρατηγική έω το 2012. Η καινοτομία αναφέρθηκε επίσης από διάφορους από τους παρεμβαίνοντες, η επιστήμη, οι επιστήμες του κλίματος συγκεκριμένα, καθώς και οι λύσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα προσαρμογής. Νομίζουμε ότι μια συνολική πολιτική ευρωπαϊκή θα μπορέσει να δώσει με την προστιθέμενη αξία τις αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα των κλιματικών αλλαγών αναπτύσσουμε το μηχανισμό του clearing house και σημειώνω και στην γνωμοδότηση του κυρίου Πρόντι την προειδοποίηση να μην έχουμε επικάλυψη προσπαθειών. Να μην επαναλάβουμε δηλαδή το σχεδιασμό συστημάτων που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν. Η άποψη τη Επιτροπή σχετικά είναι ότι χρειάζεται ο μηχανισμό clearing house για να είμαστε βέβαιοι ότι οι πληροφορίε φτάνουν από τα χέρια αυτών που τι κατέχουν στα αυτιά αυτών που χρειάζεται να τις μάθουν. Ε, εδώ έχουμε κάτι μέλη με τα δικά τους συστήματα συγκέντρωσης πληροφοριών που ήδη λειτουργούν, αλλά κάποια άλλα που δεν τα διαθέτουν καν. Τώρα, οι αναπτυσσόμενες χώρε και τα προβλήματά τους αναφέρθηκαν. Δεν ήταν αυτό το βασικό σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η Λευκή Δίβλος, αλλά αυτό καλύπτεται κατά κύριο λόγο από την ανακοίνωση πριν από τη Σύνοδο της Κομεχάγης Και βεβαίως τα όσα επακολούθησαν. Ξέρετε τι συζητήθηκε εκεί για τα 2,4 δις ευρώ και για την ε, όλη συζήτηση για την προσαρμογή. Αναφέρθηκε ανάγκη να συμπεριληφθεί η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε μια περιβαλλοντική μελέτη εντυκτύπου. Από τη δική μας την πλευρά να πω ότι θα το σκεφτούμε βεβαίω, αλλά να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Α πούμε ότι θέλετε να κατασκευάσετε ένα φράγμα. Ένα φράγμα που χρειάζεται να γίνει περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. Εφόσον όμω κανεί αποφασίσει να κατασκευάσει ένα φράγμα, έχει αποφασίσει και την τοποθεσία στην οποία θα χτιστεί το φράγμα. Οι κλιματικέ αλλαγέ λοιπόν είναι από τα σκέλη του... μια περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου, αλλά το άλλο σκέλο θα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό νερό. Δεν μπορεί λοιπόν να σκεφτούμε να οικοδομήσουμε ένα φράγμα σε ένα σημείο που δεν θα υπάρχει του άλλου νερό σε 40-50 χρόνια. Υπάρχει και το θέμα λοιπόν τη μελέτη σκοπιμότητα πριν ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξουν προγράμματα, σχεδιασμός και υποδομές για την προστασία από τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη Λευκή Βίβλο. Επίσης αναφέρθηκαν οι ζωονόσοι εδώ να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα από τα έγγραφα που συνόδευσαν τη Λευκή Βίβλο. Για την υγεία και την ευζοία των φυτών. Οι ζώνος, καλύπτονται σε αυτό το έγγραφο. Είναι ένας από τους τομείς όπου έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση η Επιτροπή. Υπήρξε πρόταση για Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προσαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι κάπως πρόημο στο στάδιο αυτό να αποφασίσουμε εάν χρειαζόμαστε ή όχι οδηγία. Επίσης έγιναν πολλές παρατηρήσεις για τη χρηματοδότηση. Η δίβλος αυτή θεωρεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σύνταξής της ούτω ή άλλω και κάπω έτσι το χειριζόμαστε το θέμα αυτό, η και κάπως ήταν ένα κινούμενο ένας κινούμενος στόχος. Θα μπορούσαμε, όπω προτείνει η Λευκή Βίβλο, να χρησιμοποιήσουμε τα εισοδήματα του ETS για την προσαρμογή στι ε, κλιματικέ αλλαγέ. Υπάρχουν ήδη κάποιε διευθετήσει χρηματοδότηση που λειτουργούν, αλλά σαφώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη χρηματοδότηση και στα πλαίσια τη αναθεώρηση του προπολογισμού των δημοσιονομικών προοπτικών. Όμω το θέμα αυτό δεν το αναπτύξαμε επαρκώ στην βίβλο, στη Λευκή Βίβλο, όπω την ενέκρινε το κολέγιο των Επιτρόπων, διότι δεν ήθελε το κολέγιο σε αυτή τη φάση να προκαταλάβει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του προπολογισμού ή για το σχεδιασμό των δημοσιονομικών προοπτικών. Δεν ήθελε να προκαταλάβει το καθεστώ χρηματοδότηση τη προσαρμογή. Υπάρχει λοιπόν περαιτέρω ευκαιρία εδώ να επανέλθουμε στο ζήτημα, να συνεισφέρετε και εσεί τι απόψει σα και να ενισχύσετε στην προσπάθειά τη στην Επιτροπή. Επίση, υπήρξαν σχέδια, προτάσεις μάλλον για το πρόγραμμα ανάκαμψη. Εδώ προτείνεται τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη την ανάγκη για προσαρμογή κατά την υλοποίηση του προγράμματος ανάκαμψης. Εδώ και οι προτάσεις για την Ευρώπη επί είναι κάτι που έρχεται να συμπληρώσει την το όλο μας σκεπτικό. Και η ανάγκη για ε, ορθολογισμό των προσπαθειών, για ευθυγράμμιση, mainstreaming, είναι κάτι που ήδη το έχουμε υπόψη. Ο πρόεδρος Μπαρόζου έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα υπάρξει μια μείζον ε, αναθεώρηση όλων των πολιτικών για να εξετάσουμε το κατά πόσο είναι εύρωστες και σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές και στο πλαίσιο που απαιτούνται, απαιτείται η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Έτσι θα αποτιμήσουμε τις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Peter Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πετρακάμελτοφ για τη θέση που μας δώσατε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δώνουμε το λόγο στον Βιτόριο Πρόντι. Να είστε σύντομο όμω, γιατί δεν μα μένει πολύ χρόνο για, για το επόμενο σημείο τη μέση διάταξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαφώς δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ε, προτάσεις που μου έγιναν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. Θα λάβω τη συνεισφορά τους υπόψη και σε πολύ συγκεκριμένα και πιο διεξοδικά θέματα. Καταρχάς, να πω το εξή Μέχρι τώρα, στην προστασία του εδάφους, το σκεπτικό ήταν πάντα να διώχνουμε τα όμβρια ύδατα το συντομότερο δυνατόν. Με την αλλαγή του κλίματος και επειδή είναι μεγαλύτερη η ένταση των βροχοπτώσεων και μεγαλύτερη διάρκεια της περίοδου ξηρασίας, θα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία μας και να προσπαθούμε να κατακρατήσουμε τα ύδατα όσο το δυνατόν περισσότερο στο σημείο στο οποίο πέφτουν. Έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη διάβρωση του εδάφους και επιτρέπουμε να ε, ξαναγεμίσουν ε, οι υπόγειες ε, υδροφόρες ε, λεκάνες οι οποίες ε, πάντα αποτελούσαν ένα μηχανισμό για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο ε, νερό και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάθε τετραγωνικό μέτρο του εδάφους προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό. Είναι κάτι βέβαια το οποίο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει μόνο εάν μαζί με το θέμα της προστασίας του εδάφου έχουμε και ανάκτηση και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, αναφέρομαι καταρχάς στην ε, συλλογή καταλήπων βιομάζας και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και τις ροές των υδάτων. Να απαντήσω εδώ και στο συνάδελφο Ρώση. Εγώ αναφέρομαι στην αύξηση της κατακράτησης του ποσοστού του ύδατος που θεωρούμε ότι θα μπορέσει να προστατεύσει από τα ξαφνικές και καταστρεπτικές συνέπειες. Εγώ λοιπόν θα ζητήσω να υπάρχει ένα σύστημα τέτοιο, ώστε να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο θέμα της προστασίας του εδάφους, η οποία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος και να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που είναι απαραίτητη για αυτή την ε, αντιμετώπιση. Έγιναν κάποιες πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις, κυρίως για τη συμμετοχή του ασφαλιστικού κλάδου. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία μεταβάλλεται ε, ταχύτατα ο κίνδυνος και οι ασφαλιστικές εταιρείε δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν αυτούς τους κινδύνους. Επομένως, για να μπορέσει να υπάρξει στήριξη του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που προκύπτουν από τις καταστροφές, θα πρέπει να υπάρξει μία συνεργασία τουλάχιστον για να μπορέσουμε να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο ε, αυτό βέβαια είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να επανέλθουμε. Είναι σαφές ότι τμήμα των πόρων θα πρέπει να προέλθει και από το μηχανισμό της εμπορίας εκπομπών, του ETS, και σαφώς εμείς θα πρέπει να επαγρυπνούμε για να μην ε, υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας και να μην ξεχνάμε ότι η κερδοσκοπία ήταν αυτή η οποία δολοφόνησε τελικά την οικονομία. Όσοι συμμετέχουν λοιπόν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών θα πρέπει ε, να ενδιαφέρονται για την ουσία και να μην ε, συμμετέχουν απλώς και μόνον ε, για να, με σκοπό το κέρδος. Ε, προσφάτως στις ε, τράπεζες υπάρχει μια συγκεκριμένη ρήτρα που έχει τεθεί ακριβώς για να βρεθούν αυτές οι κερδοσκοπικές συναλλαγές. Ε, θα σταματήσω τώρα εδώ. δεν έχω χρόνο γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο σημείο όπως μας είπατε, αλλά έχω σημειώσει όλα όσα μου είπατε και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όλες αυτές τις παρατηρήσεις στην πρόταση κειμένου την οποία θα κάνω στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε το Βιτόριο Πρόντι. Πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος είναι ένα τόσο ευρύ θέμα και σαφώς πρέπει να μας απασχολήσει εντατικά και να το προετοιμάσουμε. 12 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών για να στην, να περάσουμε στη συζήτηση στη του Μαρτίου. Το επόμενο σημείο είναι ο απολογισμός της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπενχάγη. Ήδη έχουμε συζητήσει στην Ολομέλεια για το περιεχόμενο και για τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης. Την έκθεση που προετοίμασε η Γραμματεία την έχετε λάβει. Και ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μπορώ να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε μεγάλη δέσμευση για αυτή τη διάσκεψη των ΗΕ. Ε, επισήμως είχαμε 15 μέλη, ενώ είχαμε τελικά 75 μέλη στην αντιπροσωπεία μας που συμμετέσχουν κατά τις ε, δύο εβδομάδες στην Κοπενχάγη. Και έλαβαν μέρος σε πάρα πολλές συναντήσεις, ε, συζητήσεις κλπ. Είναι πραγματικά πολύ θετικό ότι άδειξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέσχουμε σε τόσο πολλές συζητήσεις και συναντήσεις. Και γι' αυτό είναι και μεγαλύτερη η απογοήτευσή μας που τελικά δεν καταλήξαμε σε κάτι το πιο θετικό. Είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία η γραμματεία και εμείς ε, είχαμε ε, σαφώς ε, προνόμια στην πρόσβασή μας στο κέντρο γιατί δεν ήταν πολύ καλή η διαδικασία διαπίστευση ε, των δανών επιτόπου και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε και ένα συγκεκριμένο χώρο που ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το γραφείο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κοπενχάγη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο που μα διέθεσε χώρου ε, στην Κοπενχάγη. έγινε και μια συνάντηση συντονισμού Επιτροπής και Συμβουλίου όπου δεν συμμετέσχομεν και αυτό ήταν μια απογοήτευση για μας. Δεν το δέχτηκαν να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτά τα οποία θα ζητήσουμε για την διοργανική συμφωνία πριν δώσουμε την αποδοχή μας στην Επιτροπή Μπαρόζο. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες λοιπόν πρέπει να διαλευκανθεί αυτό το θέμα για το μέλλον. Μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο έχει μια θέση που έχει ενδυναμωθεί και θα πρέπει να μην είμαστε δεύτερης κατηγορίας, αλλά να μας αντιμετωπίζουν σε ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο. Είχαμε ένα πλήρες πρόγραμμα στην Κοπεχάγη. Κάθε μέρα δηλαδή υπήρχαν πολλές συναντήσεις, στις οποίες συμμετέσχομαι Πολύ ενδιαφέρουσες βρήκα τις διμερείς συναντήσεις μας ε, με διάφορα κοινοβούλια άλλων χωρών. Κίνα, Ινδία, ε, Αφρικανική Ένωση, νησιωτικέ χώρες. Ε, τι να πρωτοαναφέρω, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι συναντήσεις μας αυτές οι διμερείς. Επίσης, πολύ καλή ιδέα ήταν και οι ομάδες εργασίας, γιατί τα διάφορα θέματα που θεωρούνται σημαντικά μπόρεσαν να συζητηθούν εις βάθος της ομάδας εργασίας. Είχαμε πολλές δυσκολίες όσον αφορά τον τύπο, πολύ, πολύ αυτή η συνάντηση. Και στο ε, κέντρο που γίνονταν οι συναντήσεις δεν ήταν εύκολο ε, να βγάλει κανείς άκρη που ήταν ο τύπος που είμαστε. τέλο πάντων, όσον αφορά ε, τα μέσα ενημέρωσης, ίσως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ε, εμφάνισή μας. Δεν θέλω όμω να μονοπολίσω εγώ την παρουσίαση. Ο Καλχάινς Φλόρενς που ήταν ο αντιπρόεδρος θα μπορέσει να σας πει περισσότερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως να χρειαστεί και να επαναλάβω κάποια σημεία, αλλά ε, ε, το κύριο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της Επιτροπής που κατέθεσαν δυνατό το αδύνατον πραγματικά. 70 βουλευτές να τους χειριστούν, να τους ε, κατευθύνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, ε, τα μέλη της Γραμματείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια γιατί καταφέρατε να φροντίσετε τα πάντα. Έχω πάει σε πολλές συναντήσεις και έχουμε δει πώς ε, οργανώνονται αυτές οι πολυμερείς ε, συζητήσεις και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας. από τα 15 μέλη στο Μπαλί φτάσαμε τώρα στα 73 και καταλαβαίνει κανείς γιατί είχε και τεράστια οργανωτικά προβλήματα αυτή η συνάντηση και τίθεται και το θέμα αν πραγματικά είναι, διαπραγμα... αν πραγματικά είναι διαχειρίσιμο ένα τόσο μεγάλο μέγεθος ε, συναντήσεων. Είναι τα πάντα γεμάτα, είναι τα πάντα ε, παραφορτωμένα. Αυτά για τα οργανωτικά. Την περίπτωση εβδομάδα δεν μπορούσα να είμαι στο Στρασβούργο για να συζητήσω αυτά τα θέματα. Το αποτέλεσμα σαφώς ε, δείχνει κάποιες αδυναμίες. Ε, δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε. Μια κάποια επιτυχία θα μπορούσαμε ε, να πούμε ότι είχε η διεξαγωγή αυτή τη συνάντηση. Ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπιών. Γιατί αν συναντιόντουσαν τρει αντιπροσωπείε, άλλε τρει αντιπροσωπείε κάπου αλλού θεωρούνταν ότι αποκλείστηκαν και καθόντουσαν στη γωνιά τους παραπονούμενες. Ε, δεν είχε ζωή δηλαδή αυτή η συνάντηση της Κοπενχάγης όπως θα τη θέλαμε. Ε, αυτό ισχύει και για τη συνάντηση των επικεφαλής κρατών. Αυτό το οποίο θεωρούμε καλό για την Ευρώπη, μάθαμε ότι δεν είναι αναγκαστικά καλό και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν πολλές διαφοροποιημένες δράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. και πρέπει να σκεφτούμε αν ε, πρέπει να συνεχίσουμε πάνω στα ίδια πράγματα που συζητούσαμε μέχρι τώρα, ή πώς πρέπει να σκεφτούμε και νέους τομείς που πρέπει να συζητηθούν. Ευχαριστώ. Στο συμπρόεδρο δώσαμε ένα λεπτό παραπάνω, λοιπόν. Δίνω το λόγο στη Λίντα Μακάβαν τώρα. Um, Δύο λεπτά. Να ευχαριστήσω ξανά, ιδίω την Γραμματεία, για την εξαιρετική τη δουλειά και κυρίως που μας βοήθησε να έχουμε πρόσβαση στα διάφορα κτίρια με τόση αποτελεσματικότητα κάποιες φορές. Είχαμε σαφώς ε, καλή εικόνα των διαπραγματεύσεων που έγιναν σε διάφορα επίπεδα. Αυτό που τώρα μας ανησυχεί είναι τι θα γίνει με τη νέα επιτροπή όταν θα έρθει εδώ και θα χρειαστεί να μας εξηγήσει τι γίνεται μετά την Κοπενχάγη. Διότι καταλαβαίνω ότι από την 31η Ιανουαρίου, αυτό έγινε σαφές και την 5η, η προθεσμία δεν ισχύει πλέον η συμφωνία ε, σημειώθηκε βεβαίως από την ε, Σύμβαση των Μερών, όμως ε, κανείς δεν φαίνεται να δεσμεύεται από τη συμφωνία. Και αποφασίστηκε, ουσιαστικά ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη σε εσωτερικό επίπεδο να λάβουν δεσμεύσεις για τους στόχους τους, εάν θέλουν. Τίποτα το δεσμευτικό λοιπόν περί στόχων δεν αποφασίστηκε. Θέλω λοιπόν απόλυτη σαφήνεια για το ποια είναι η ευρωπαϊκή θέση αντιλαμβάνομαι ότι το Συμβούλιο μιλάει για τον στόχο του τριπλού 20. Τα κράτη-μέλη προτείνουν άλλους αριθμούς και έχει περιέλθει σύγχυση για το μετά την Κοπενχάγη στάδιο. Τι σημαίνει από νομικής άποψης αυτό που αποφασίστηκε εκεί, τι θα γίνει μετά. Εγώ πιστεύω ότι πολλά έχουν χαθεί στον δρόμο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πολύ προσεκτική παρακολούθηση του θέματος για να έχουμε επιτελέσει πρόοδο στο τέλος της χρονιάς. Ευχαριστούμε κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και εσάς τον ίδιο για τα όσα κάνατε σε αυτή τη σύνοδο. Πάντως, ως βουλευτές, δεν μπορούμε να άκρος απογοητευμένοι. Τελείως απογοητευμένοι από την θέση που είχε επιφυλαχθεί στο Ευρωκοινοβούλιο στην όλη διοργάνωση της Συνόδου. Δεν υπήρχε πραγματικά θέση στο πλευρό του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Βεβαίως κάθε πρωί είχαμε μία απενημέρωση, αλλά ήταν απλώς ενημερωτική η συνάντηση αυτή, δεν πρόκειται για πρόσκληση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και συμβολικώς να πω ότι δεν υπήρχαν καν τα badge που θα μας επέτρεπαν την πρόσβαση στην Ολομέλεια οι κάρτες δηλαδή πρόσβασης. Ε, κάτι πολύ μικρό αλλά συμβολικότατο. Μόνο κάποια περιορισμένα μπάτζ υπήρχαν για τον κύριο Λόρεν, εσά, τα οποία έπρεπε να τα ανταλλάσσετε και μεταξύ σα. Πάντω, δεν προβλεπόταν να επίσημη συμμετοχή των μελών του Ευρωκοινοβουλίου στη Συνόδο τη Ολομέλεια. Εγώ, μάλιστα, έγινα μάρτυρα ε, αυτού του γεγονότος. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με τη δική σας διοργάνωση, την ε, πλευρά του Κοινοβουλίου, αλλά το πώς ε, το μεταχειρίστηκαν το Κοινοβούλιο σε αυτή τη σύνοδο της Κοπενχάκης. Κατά τα άλλα, σαφώς συζητήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, ε, είχαμε ευκαιρία στα, στις διάφορες εκδηλώσεις στο περιθώριο να συζητήσουμε πολλά από τα συμμετέχοντα μέρη, αλλά η συμμετοχή μας δεν ήταν ενεργή. Δεν μπορεί κανείς να πει, νομίζω, ότι συμμετείχε πραγματικά στην μία στην άλλη συζήτηση. Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται κυρίω στη γραμματεία που μας προετοίμασε τη συνάντηση. Και ήταν ενδιαφέρουσε συναντήσει με τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα τα κοινοβούλια στο μέλλον. Ήταν μεγάλη η βαρύτητα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων αυτή τη φορά. Θα του χάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, συμφωνώ με όσους ε, εξήμνησαν το έργο της Γραμματείας. Ευχαριστώ και εκ μέρους μου στη Γραμματεία. Το θέμα της διαπίστευσης τώρα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, δεν είναι βέβαια κατά πόσον ε, θα μπορούν ε, να συμμετάσχουν και αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει μια νέα διαπραγμάτευση, μια νέα συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε κάθε το μέλος να έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα διαπίστευσης μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλο τώρα το να υπάρχουν περισσότερα μέλη και να υπάρχει πρόσβαση για όλους ε, στις διάφορες συνεδριάσεις που γίνονται. Αλλά τουλάχιστον το θέμα της διαπίστευσης στην είσοδο θα πρέπει να δίνεται σε όλα τα μέλη. Δεύτερον, Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία θα πρέπει να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι χρειαζόμαστε μια πιο δραστήρια πολιτική για το κλίμα. Δεν αρκεί το να έχουμε εξαιρετικού εμπειρογνώμονε που να γνωρίζουν την κάθε λεπτομέρεια αυτή της διαπραγμάτευση. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη προσπάθεια για την διπλωματία και όλα σε θέματα κλίματος να μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις βασικές ε, χώρες λεγόμενες, οι οποίες φάνηκαν να είναι πιο δραστήριες ε, στα θέματα του κλίματος από ό,τι στο παρελθόν και διαδραμάτισαν και πολύ ουσιαστικό ρόλο στα όσα διαμήφθησαν στην ε, Κοπενχάγη. Πολλοί έθεσαν ερωτήσεις για το κατά πόσον η Κίνα που ανήκει σε αυτή την ομάδα βασικών χωρών βρίσκονταν πίσω από το Σουδάν για να μην, υπάρχει, να μην υπάρξει τελικά η συμφωνία στην Κοπενχάγη και να μην έχουμε επίσημη απόφαση. Μια τρίτη παρατήρηση. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να βρει τρόπους να μην σταματά η διαδικασία διαπραγμάτευσης, να υπάρχει μια απόφαση στα Ηνωμόνα Έθνη, ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον ε, κάποιοι κανόνες, κυρίως σε διαδικαστικά θέματα, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες. Thank you very much. Ε, η κυρία Ντεμπρούν, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με όλους όσους ε, είπαν ε, για το ότι σημειώθηκε η συμφωνία, ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη Διεθνή Συμφωνία το 2010 και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι κυρίως ε, όσον αφορά στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι στόχο θα πρέπει να έχουμε εμείς, δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο ένα 20%. Στην Ολομέλεια κάποιοι ζήτησαν 30%, εγώ ζήτησα 40%, αλλά νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να βρούμε νέους τρόπους, ώστε να είμαστε συνεχώς ε, δραστηριοποιημένοι στο θέμα αυτό και να δούμε και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις με τους ε, άλλους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Γραμματεία που έκανε εξαιρετική δουλειά και μάλιστα υπό δύσκολε συνθήκε και να ευχαριστήσω και εσά κύριε Πρόεδρε και την Task Force ε, και ε, με όλου όσου συμμετείχαν στο τμήμα επικοινωνία. Ε, νομίζω ότι κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όσον αφορά στο θέμα της πρόσβασης, Νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να γράψουμε μία επιστολή η οποία θα απευθύνεται σε όλους όσους οργανώνουν ε, το θέμα και από πλευράς Δανίας και από πλευράς Ηνωμένων Εθνών για τη διαδικασία διαπίστευσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επίσημη διαμαρτυρία του θέματος και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τις δικές μας εσωτερικές διαδικασίες. Ποιο συμμετέχει σε μια αντιπροσωπεία, ποιο δεν συμμετέχει, ώστε να είναι λίγο πιο σαφή τα πράγματα εκ των προτέρων για όλους όσους σκοπεύουν να μεταβούν εκεί ε, και τι δυνατότητες θα έχουν. Νομίζω ότι κάποια από αυτά και σε εμά ε, σαν αντιπροσωπεία έρθαν λίγο καθυστερημένα. Και επίσης να πω ότι υποστηρίζω και τις μελλοντικέ διαδικασίες. Να συνεχίσουμε δηλαδή να ζητάμε πρόσβαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορεί να συμμετέχει και στις συντονιστικές συνεδριάσεις. Ευχαριστούμε. Άννα Ρότσμπαχ. Yeah. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τη γραμματεία για όσα έκανε στη Σύνοδο της Κοπεχάγης. Πολύ καλά τα οργάνωσε. Εγώ είμαι Δανέζα. Οπότε η θέση μου είναι κάπως δύσκολη. Δεν μπορώ να, παρα... να παραδεχτώ ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα. Αλλά Σίγουρα κάπως με ενόχλησε όταν είδα τους συναδέλφους μου να μένουν ώρες και ώρες στο κρύο περιμένοντας να καταφέρουν να μπουν στο κέντρο της των συνεδριάσεων. Πραγματικά και εγώ ίδια δεν μπορώ να δικαιολογήσω τα όσα συνέβησαν. Το συζήτησα με διάφορους υπευθύνους και φαίνεται ότι δεν υπήρχαν παρά μόνο τέσσερις κάρτες πρόσβασης, τέσσερα μπάντζ. Γι' αυτό η αίθουσα ήταν μισοάδια και αυτό ήταν αρκετά ενοχλητικό δεν το είχαμε μάθει ότι δεν θα είχαμε παρά μόνο τέσσερις κάρτες στη διάθεσή μας, ενώ το κέντρο θα έμενε άδειο. Δεν έπρεπε λοιπόν να έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, αυτό είναι σαφές. Και σίγουρα για την επόμενη φορά θα πρέπει από πρακτική άποψη να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Συμφωνώ απολύτω πάντω ότι οι συνάδελφοι που θέλουν να εκφράσουν επισήμω ε, τη δυσαρέσκειά του να το κάνουν και εγώ θα συνυπογράψω μαζί του. Έχουν δίκιο. Πάντω να πω ειλικρινώ ότι δεν είχα και φοβερέ προσδοκίε από αυτή τη σύνοδο. Είχαμε θέσει τον πύχη αρκετά ψηλά και είναι η πρώτη φορά που τόσε πολλέ χώρε συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν ένα ζήτημα που αφορά όλου. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τόσα διαφορετικά επίπεδα από άποψη οικονομική, γεωγραφική, πολιτιστική. Εγώ ήλπιζα ότι θα καταλήγαμε σε κάποιο είδους σχέδιο σχεδίου συμφωνίας, ότι θα είχαμε ένα έγγραφο που θα ήταν μια βάση, ένα σημείο αφετηρίας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον τις συζητήσει. Αυτά τα βασικά θεμέλια για το αρχιτεκτόνημά μας, ε, για να συνεχίσουμε στο Μεξικό όχι, δεν ξέρω αν να τα έχουμε. Σίγουρα το μετρό λειτουργούσε και αυτό είναι σαφώς υποδομές. Νικ Γκρίφιν. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εγώ τη Γραμματεία. Η συνάντηση COP15 νομίζω είναι μια συνάντηση στην οποία εμείς συζητούσαμε για αυτά τα οποία συζητούσαν κάποιοι άλλοι. Πλήρη κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Εν πάση περιπτώσει, για να είμαι θετικό, να εκφράσω κάτι θετικά, πρέπει να πω ότι υπήρχε μια γερμανική εταιρεία με τεχνολογία ε, που ε, αφορά ε, κράματα άνθρακα που θα είναι πολύ πιο ισχυρό από τον ανοξίδωτο άνθρακα, τον ανοξίδωτο χάλιβα συγγνώμη, και πολύ πιο ανθεκτικό από το τσιμέντο και ε, ήταν μια τεχνολογία πολύ χρήσιμη που μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να μειώσει τον κινέζικο χάλιβα, παραδείγματο χάρη που χρειαζόμαστε. Και υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε να βοηθήσουμε τον τρίτο κόσμο με φτηνέ κατοικίε που δεν θα χρειάζονται τη χρήση ξύλου ε, πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία. Θα ενημερώσω την Επιτροπή αν θέλετε και δεν ξέρω αν και οι άλλοι παρευρισκόμενοι είδαν αυτή την τεχνολογία. Είναι κάτι θετικό που μπορούμε να φέρουμε από την Κοπενχάγη γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι φαντασιώσεις για το κλίμα. Ας δούμε λοιπόν κάτι συγκεκριμένο που θα βοηθήσει τους ανθρώπους και στην Ευρώπη και τους φτωχού ολόκληρο τον κόσμο. Άρα δεν ήταν εντελώ περί τη Κοπενχάγη, βρέθηκε και μια καινούργια τεχνολογία στην Κοπενχάγη. Ο κύριος Κυλακάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πήγα στο Μπαλί και στο Πόσναν και συμμετείχα και στις ε, διαπραγματεύσεις της δικής μου κυβέρνησης και από την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου αυτό το οποίο πήρα ήταν πολύ καλύτερο. Και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς που το οργάνωσαν. Μπαίνοντας τώρα περισσότερο στα αποτελέσματα της διάσκεψης, θα πω τα Νομίζω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τη στρατηγική μας. Μου έκανε εντύπωση πόσο αδύναμη ήταν η θέση μας όταν συζητούσαμε με τις αντιπροσωπείες της Κίνας και της Ινδίας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ε, οι Κινέζοι πήραν ένα ποτήρι και είπαν έχουμε 30 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν πίνουν τέτοιο χρώμα νερό, αλλά τέτοιο χρώμα νερό, αυτό ήταν μια στιγμή που στο μυαλό μου το όλο θέμα της Κοπενχάγης ένιωσα ότι έληξε. Δεν είχαμε επιχειρήματα έναντι των Κινέζων όταν μιλούσαν ε, για τις δικές τους θέσεις. Κάτι το οποίο και η Ινδία εξέφρασε με κάπως πιο ήπιο τρόπο. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέα στρατηγική και νέα επιχειρήματα σε αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχουν νέα επιχειρήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Παραδείγματο χάρη, ορυκτά καύσιμα. Δεν τα συζητήσαμε. Δεν συζητήσαμε το θέμα των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, που είναι μια πολιτική τεράστια σημασία στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα Μιλάμε για αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα. Και πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για μια προοπτική ευρύτερη, για το 2050 ενδεχομένως, όταν οι Κινέζοι και οι Ινδοί θα έχουν παρόμοιες ευθύνες, συγκρίσιμες. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Euh, Πρόεδρε, λίγα λόγια αφού ευχαριστήσω και εγώ τη Γραμματεία για την πολύ καλή διοργάνωση μας υποδέχτηκαν με πολύ καλό τρόπο. Μπορέσαμε να δούμε και πώς άλλοι προσκεκλημένοι έγιναν δεκτοί γιατί βρισκόμασταν στο ίδιο ξενοδοχείο. Ε, σίγουρα απομένει κάποια πρόοδο που θα μπορούσε να γίνει, Πρόεδρε. Τέλος πάντων, για να σοβαρευτώ και λίγο. Στην Κοπενχάγη τρία πράγματα μας έμειναν. Ε, μια, ένα παράπονο και μια ελπίδα Και επίσης, όπως έλεγα προηγουμένως και όπως έλεγε η κυρία Λεπάζ, το παράπονο μας είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε αρκετά σε αυτή τη συζήτηση. Η απουσία του έγινε αισθητή τις τελευταίες ώρες λόγω των ε, διαφωνιών που υπήρξαν ήδη στα πλαίσια της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής. Δεν φανήκαμε στο ύψος των περιστάσεων δυστυχώς και εμείς που από την πλευρά του Κοινοβουλίου μεταφέραμε την αποφασιστικότητά μας να βρούμε μια συμβαστική λύση, μπορούμε να είμαστε απογοητευμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να είναι ένας ενεργός παράγοντας στις συζητήσεις της Κοπενχάγης. Το παράπονο λοιπόν είναι ότι εμείς οι ίδιοι μείναμε θεατές των εξελίξεων. Παρόλα που με τη διοργάνωση συναντήσεων των διαφόρων αντιπροσωπιών μπορέσαμε διαζώσεις να δούμε τις δυσκολίες που ενέχουν τέτοιες διαπραγματεύσεις. Και η ελπίδα μας, αυτό που ήθελα να πω για να κλείσω, είναι ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης ενδεχομένως για τέτοιου είδους συνόδους. Ίσως εμείς να μπορούμε να κάνουμε προτάσεις. Ευχαριστούμε κύριος Έικουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Βεβαίως θα ευχαριστήσουμε τη Γραμματεία για τον προγραμματισμό εγώ ήμουν σε στενή επαφή με του πράσινου συναδέλφου από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο και ομολογώ ότι εκείνοι ξαφνιάστηκαν με το δικό μα πρόγραμμα σε σχέση με το δικό του. Η γραμματεία μα τα οργάνωσε πολύ καλά. Για την Κοπεχάγη δεν θέλω να συζητήσω τώρα, θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε πιστεύω στο μέλλον. Όμω, αυτό που θέλω να προσθέσω στι προηγούμενε παρατηρήσει είναι ότι ω κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί με τον εαυτό μα. Δηλαδή, καταβάλαμε μεγάλε προσπάθειε για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση του Ευρωκοινοβουλίου με το ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο, αλλά τελικά η απόφαση αυτή που εκφράζει την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ούτε που αναφέρθηκε το Δεκέμβριο. Λοιπόν, η θέση για την οποία τόσο μοχθήσαμε προκειμένου την αποσπάσουμε, το θέμα είναι πώς θα βελτιωθεί. Είναι σημαντικό, πιστεύαμε, αλλά σχεδόν ούτε ασχολήθηκε κανείς, ακόμη και στις ενημερώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε άλλε δηλώσει έδιναν και εκείνη η έμφαση, οι οποίε δεν είχαν και καμία σχέση με τα όσα εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο είχαμε συμφωνήσει. Εμεί λοιπόν ω βουλευτέ πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι όταν δεν ακολουθείται η θέση μα, αυτό θα πρέπει να μα απασχολεί. Αλλιώ να διερωτώμεθα γιατί κάνουμε αυτά τα ψηφίσματα, γιατί τα ετοιμάζουμε, γιατί ετοιμάζουμε τι αποφάσει. Μόνο για να ξοδεύουμε χαρτί και μετά να πηγαίνουμε στην Κοπενχάγη και να συζητάμε θεωρητικά, χωρί να θίγεται καν η θέση μα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πιο αυστηροί με τον εαυτό μα, όπω και με την Επιτροπή ζητάμε να είναι πιο συνεπεί στι υποχρεώσει τη. Να βελτιώσουμε λοιπόν τη θέση μας την ίδια στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Παίζουμε ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς, αλλά στα Ηνωμένα Έθνη δεν παίζουμε ρόλο. Αυτό είδαμε στην Κοπενχάγη. Ο Βιτόριο. <coughs> Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να προσθέσω και εγώ τις ευχαριστίες μου, τις θερμές μου ευχαριστίες στο προσωπικό διότι αισθανθήκαμε πραγματικά ότι το πρόγραμμα ήταν πολύ καλό. Βεβαίω υπήρξε τεράστια απογοήτευση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε σε κατοπινό στάδιο, αλλά να πω ότι αυτό που κυρίως έλειπε ήταν μια απόκριση στα... και η συνέχεια του Μπαλί. Και μια αίσθηση κοινή ευθύνη. Γι' αυτό δεν είχαμε προετοιμαστεί. Δηλαδή, εγώ είχα προσπαθήσει επανειλημμένως να προτείνω τη συμπερίληψη των ρητρών ισότητας και ισοδυναμίας στην όλη συζήτηση και δεν τα είχα καταφέρει. Η ήττα που γνωρίσαμε, η έλλειψη αποτελεσμάτων από την Κοπενχάγη μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τελείως στάση. Η πρότασή μας έτσι όπως ήταν διαθρωμένη ήταν αρκετά περιορισμένη. Αλλά τελικά γι' αυτό και οδήγησε στην απομόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον αποκλεισμό της από την τελική συζήτηση. Εφόσον ήταν πολύ συγκεκριμένη στη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπόλοιποι τα βρήκαν μεταξύ τους και μας μας έβαλαν στην άκρη. Αυτό συνέβη. Είναι τελείως παράδοξο βέβαια αυτό, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε στο μέλλον τις προτάσεις μας, να τις έχουμε προετοιμάσει επαρκώ, να είναι τελείω διαφορετικέ. και να έχουμε από την αρχή σκεφτεί την ανάγκη πολιτικής ε, έκβασης και επίλυσης των όσων προβλημάτων είχαν τεθεί και στον Παλί. Ευχαριστούμε. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Ορέστε Ρώση. Ναι, συμφωνώ απολύτως και εκτιμώ τα όσα είπε ο συνάδελφος Πρόντι. Αντιληφθήκαμε όλοι ότι το να ζητάμε πολλά και να παρουσιάζουμε ένα υπερβολικό ψήφισμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ε, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, συγγνώμη, μπορούσε και τελικά οδήγησε σε πάυση των συζητήσεων. Πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι, να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε για το COP16, για την ε, Κοπεχάγη 16 και να είμαστε ήδη έτοιμοι. Να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε με τη ΣΥΠΑ, την Ινδία, την Κίνα, την Αφρική, ε, δυνάμεις ε, λίγο πολύ στεναρές, οι οποίες όμως δεν θα δεχθούν ποτέ πράγματα σαν αυτά που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι απίστευτο κύριε Πρόεδρε, αλλά για πρώτη φορά συμφωνώ μαζί σας. Με η Κομπεχάγη 15 δεν ήταν επιτυχία, αλλά συμφωνώ μαζί σας για την επιστολή διαμαρτυρίας, είτε γραπτή είτε προφορική τέλος πάντων, ε, ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε εμείς είμαστε υπέρ. μετά από τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ερχόμαστε μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο. Οι εκπρόσωποι μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιμένουν στο δρόμο ή έξω από μια αίθουσα. Αυτό αποτελεί προσβολή για τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το ίδιο το θεσμικό όργανο. Ε, είναι ευπρόσδεκτες λοιπόν οι διαμαρτυρίες σας, με χαροποιεί ιδιαίτερος και εύχομαι να υπάρχει και κάτι επί χάρτου. Επαναλαμβάνω, ε, συμφωνώ και πρέπει να αποσταλεί σε όλους τους οργανισμούς και σε όλα τα θεσμικά όργανα. Εύχομαι να είναι μεγαλύτερη συνεργασία για την Κοπεχάγη 16 και να έχουμε και ένα έγγραφο το οποίο ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει και τη βάση επί της οποίας θα ξαναγραφτούν οι μελλοντικέ αποφάσεις ε, ε, στα θέματα του κλίματος. Άλλοι δύο μιλητές. Ε, Μιχαήλ Τρεμόπουλος και Γιώργος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Σαν επιπρόσθετα σε αυτά τα οποία ακούστηκαν ως κριτική, εγώ θα πω κάτι παραπάνω. Ότι η διάσκεψη αυτή της Κοπεχάγης ήταν ένα φιάσκο. Και ακριβώς γιατί ποτέ τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν μαζεύτηκαν για να πετύχουν τόσο λίγα πράγματα. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε την πρωτοπορία που είχε ε, στον τομέα στο παρελθόν. Και φυσικά αν κρίνει κανείς από το οικολογικό αποτύπωμα όλων αυτών των ανθρώπων που μαζεύτηκαν εκεί ήταν ε, τελικά σε βάρος του κλίματος. Είπατε για 15 ε, επίσημα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου που ήταν εκεί που στην πράξη έγιναν 75. Καταλαβαίνω το ότι κάποιοι έχουν το χρέος να μας εκπροσωπήσουν σε κάποιες συνομιλίες επίσημα στις διαπραγματεύσεις. Ποιος ήταν ο ρόλος για τους άλλους 60. Υπήρξε ένα κεντρικό γεγονός που να δημιουργήσει κάποια αίσθηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωριστά από όλες τις άλλες αντιπροσωπείες. Τουλάχιστον η λίστα των συμμετεχόντων θα έπρεπε στον, απολογισμό να υπάρξει. Υπάρχει ένα οργανωτικό έλλειμμα και δεν μιλάω για αυτά που έκανε η δικιά μας γραμματεία. Μιλάω για σημαντικά οργανωτικά ελλείμματα των οικοδεσποτών ε, στην ίδια την ε, Κοπεχάγη. Και ε, βέβαια το πολιτικό έλλειμμα είναι αυτά που υπόθηκαν και ως κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν περίμενα κανέναν να μου δώσει τη δυνατότητα να μπω γιατί έχω προβλέψει. Είχα μια αντίστοιχη εμπειρία και το 2002 στο Johannesburg. Μπήκα ως εκπρόσωπος NGO και δεν έχασα στιγμή αυτά που ήθελα να παρακολουθήσω. Όμως οφείλω να σας πω ότι σημαντικά για μας είναι και αυτά που έγιναν από την κοινωνία των πολιτών. Το κλίμα φόρουμ που ήταν εξαιρετική διοργάνωση και έβγαλε επίση ένα δικό του ντοκουμέντο, αλλά και η μεγάλη διαδήλωση των 100.000 ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί και πίεσαν από όλε τι γωνιές του πλανήτη με το δικό του τρόπο για να πάρθει σοβαρά το δικό του μήνυμα. Θα ήθελα κλείνοντα για τη συνέχεια να πω ότι μπροστά μα είναι φυσικά το Μεξικό, αλλά είναι και η Βολιβία, είναι και η βόνη και θα ήθελα η δικιά μας τουλάχιστον Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες αυτές τις διεθνείς οργανώσεις που στοχεύουν στον ίδιο σκοπό για τον οποίο εμείς εδώ συζητάμε. Azt gondolom Στην Ουγγαρία λέμε κάτι το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ για να περιγράψουμε την κατάσταση στην Κοπενχάγη. Λέμε πολύ κακό για το τίποτα, με λίγα λόγια. Και νομίζω ότι αυτό ήταν αυτό που μπορεί να περιγράψει στην Κοπενχάγη. Σίγουρα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση επί των θεμάτων, γιατί μας ενδιαφέρει να έχουμε μία άποψη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει, ε, Πρόεδρε, να έχετε και να έχει και η Επιτροπή τη δυνατότητα να κάνουμε ανταλλαγές απόψεων εις βάθος και να δούμε γιατί δεν είχαμε ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έχω κάποιες ιδέες, έχω κάποια πράγματα κατά νου και σίγουρα δεν πρόκειται τώρα να σας τα θέσω όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε σε βάθος στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. θα τα προωθήσουμε στον Πρόεδρο για να τα προωθήσει και στη Δανία και στον, στα Ηνωμένα Έθνη. Και με την Νέα Επιτροπή θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για το Μεξικό στο δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, γιατί μείναμε λίγο παραπάνω στι 12.30. Θα συνεχίσουμε στις 3 με την Υπουργό Υγείας της Ισπανίας.